πέρασμος αλλά ο αριθμός των ατόμων που ήρθαν από την Νότια μέσο είναι πολύ λίγοι, ε, πολύ μικρός. Ε, δεν το ξέρει κανένα σχεδόν το πρόγραμμα έρασμος εκεί. Θα πρέπει επίσης να διαφημίσουμε αυτή τη δυνατότητα. Ε, οπότε μέγιστη ευελιξία είναι απαραίτητη. Όταν μιλάμε για προθεσμίες, για περίοδους μαθητείας, ωράρια, για τους ε, φοιτητές που βρίσκονται σε μαθητεία θα πρέπει να είναι όσο πιο ελαστικά γίνεται γιατί ε, μερικές φορές δεν έχουν νόημα οι περιορισμοί αυτοί γιατί εξαρτώνται από το ακαδημαϊκό έτος, το χρονοδιαγραμμά του, το ημερολογιό ε, ή τον τύπο μαθητείας κλπ. Οπότε θα πρέπει να είμαστε πολύ ελαστικοί. Και το πρόβλημα ουσίας είναι η απώλεια μυαλών από αυτές τις χώρες ε, και η περίπτωση δημιουργίας ενός σχήματος λαθρομετανάστευσης. Όμως το πείραμα αξίζει τον κόπο γιατί κανένας δεν θέλει να του φύγουν τα καλύτερα μυαλά και εμείς από την άλλη μεριά ενδιαφερόμαστε η μετανάστευση να γίνεται με, ε, σύμφωνα με τον νόμο και τους τύπους. Ναι, προφανές ότι ε, υπάρχει πολύ περιθώριο ακόμα γιατί για τους επιχειρηματίες και τον οικονομικό κόσμο ε, οι θεωρήσεις δικηγόρων, επιχειρηματιών, ανθρώπων οι οποίοι έχουν οικονομικές σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να εξασφαλιστεί και δεν συμπεριλαμβάνονται όλοι αυτοί στη συγκεκριμένη πρόταση. Ούτε επιχειρηματίε, ούτε δικηγόροι, ούτε τίποτα από αυτά. Πλην όμω και πάλι είναι ένα καλό ξεκίνημα. Φοιτητέ, σπουδαστές, οι ερευνητές είναι μια καλή αρχή. Γιακολίνο. Γιακολίνο. Δεν... Λοιπόν, ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα είμαι λακωνικότατος. Η οδηγία που σχολιάζεται μια οδηγία που ακολουθεί τη σωστή κατεύθυνση και πολλές πλευρές συμπληρώνει τις άλλες ε, που αφορούν την εποχιακή εργασία και άλλες. Θα πρέπει να κάνουμε διάκριση μεταξύ αυτής της οδηγίας που αφορά τους φοιτητές, τους ερευνητές και εγγυάται την πλήρη αξιολόγηση των ταλέντων, των νέων ταλέντων που προέρχονται από τίτες χώρες από τις άλλες. Χτες ο Πάπας πήγε στη Λαμπεντούσα, ο Πάπας Φραγκίσκος ήθελε να εκπροσωπήσουν τον καλύτερο τρόπο την ισχυρή αντιπαράθεση σε αυτό που αποκάλυψε την παγκοσμιοποίηση της αδιαφορίας, στρεφόμενος προς τους μετανάστες διαφορετικής θρησκείας ε, που ε, ενστερνίστηκαν αυτά που είπε. Θα πρέπει να απευθυνόμεθα προς νέους που έχουν την απέτηση εμβάθυνσης των γνώσεών τους. Είμαι πεπισμένος ότι αυτή η οδηγία, αυτή η πρόταση μπορεί να τονώσει, να δώσει κίνητρα στην Ιθωνική Προεδρία να ξεπεράσει τις δυσκολίες στις, ε, και θα ξεπεραστούν οι δυσκολίες ε, στην τελευταία φάση. Και εγώ είμαι εισηγητής ε, όσον αφορά την ICT για την κινητικότητα εντός Ευρώπης. Ελπίζω λοιπόν να ενισχυθεί αυτή η όθηση από τις συναντήσεις αυτές όπως σημερινή. όσον αφορά τις, τις τροπολογίες συγγήτριας έχω προβληματισμό. Όσον αφορά την θελοντική εργασία, τη μία αμοιβόμενη εργασία, Εκεί ε, θα ήθελα να έχω και άλλες ε, πληροφορίες. Μου είναι απαραίτητες αυτές οι πληροφορίες για τις ε, δραστηριότητες και ελπίζω ότι με την πάρα του χρόνου θα κάνω την ανάλυση. Ευχαριστώ κύριε Γιακολίνο. Είμαστε έτοιμοι για την ψηφοφορία. Ας ακούσουμε όμως μετά από όλα αυτά τα σχόλια και την εισηγήτρια. Κύριε Βίξτρομ, ευχαριστώ πολύ. Εκτιμώ πάρα πολύ όλα τα σχόλια από τους συναδέλφους ιδιαίτερα τους ε, σκιώδεις εισηγητές. Και η Ανά Μαρία Κοράτσαμπίλτ και ο Κυριακός Τριανταφυλλίδης ρώτησαν ε, το ίδιο πράγμα. Γιατί δηλαδή θέλω να παρατείνω το δικαίωμα παραμονής από 12 σε 18 μήνες και ποιο είναι το σκεπτικό πίσω από αυτό. Να σας πω λοιπόν ότι σήμερα υπάρχει, υπάρχουν πάρα πολλές ε, διαφορές στα κράτη-μέλη. Στη Σουηδία για παράδειγμα οι φοιτητέ ή ένας γιατρός που αποφυτά από το πανεπιστήμιο δεν χρειάζεται κανένα μήνα να περιμένει. Μηδέν. Στη Γερμανία είναι 18 μήνες το διάστημα αυτό. Η ενα γιατρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν 12 μήνες. Ε, όμως, ε, 18 μηνε ό,τι καταλαβαίνω, η προταση τη ευρωπαικη επιτροπη ηταν 12 μηνε ε ομως ε απο οτι επιτύχει στο να προσελκύσει τα νέα ταλέντα. Έχουν λοιπόν εκεί 18 μήνε, Γι' αυτό και εγώ πρότεινα τους 18 μήνες, διότι αφού γίνεται στη Γερμανία, γιατί να μην γίνεται και οπουδήποτε αλλού στην Ευρώπη. Οι κάτω χώρες, για παράδειγμα, έχουν κρατήσει τους 12 μήνες. Μίλησα πρόσφατα με, τον, με την πρίτανη του Πανεπιστημίου του Σουψάλα στη Σουηδία και μου είπε ότι σημασία δεν έχει ο χρόνος, αλλά η δυνατότητα παραμονής για κάποιο χρονικό διάστημα. Και ε, εντάξει δεν πιστεύω πόσο σημαντικό είναι το 12 ή το 18 το νούμερο δηλαδή. Θα βρούμε κάποιον συμβιβασμό, αλλά όπως είπα, αφού γίνεται στη Γερμανία θα γίνεται και οπουδήποτε αλλού. Αυτό είναι το σκεπτικό μου. Τώρα, συμφωνώ με τους συναδέλφους που Έφυξαν το θέμα ρύθμιση ε, τη αγορά εργασία στα κράτη-μέλη. Δεν πρέπει να ρυθμίσουμε όντω την αγορά εργασία, αλλά είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε μια ελάχιστη πρόσβαση στου φοιτητέ ε, προ την αγορά εργασία. Αυτό πρέπει να τονιστεί. Τώρα, τι άλλο. Ναι, κάποιο ανέφερε ότι αυτό ίσως είναι ένας τρόπος να αποφύγουμε τη διαρροή εγκεφάλαιων όπου τα νέα ταλέντα εγκαταλείπουν την Ευρώπη. Ναι, αυτό είναι, ακριβώς αυτό. Θέλουμε να κάνουμε κάτι για να προσελκύσουμε ταλέντα και να κρατήσουμε εδώ τους ερευνητές, τους γιατρούς, τους επιστήμονες και να μην τους ε, αναγκάσουμε να τρέξουν στις Ηνωμένε Πολιτείε ή κάπου αλλού με το που αποφυτίσουν από κάποιο ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο. Θέλουμε να μείνουν και αυτό είναι ένας πολύ καλός τρόπος να τους το δείξουμε. Επίσης, η πρίτανης του Πανεπιστημίου του Σουψάλια μου είπε ότι δεν αρκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να τους δώσει ένα πτυχίο, ένα διδακτορικό και μετά να αναγκάζονται στη Σουηδία να φύγουν μέσα σε δέκα μέρες. Εάν έχουν τη δυνατότητα να μείνουν για 12 ή για 18 μήνες, είμαι σίγουρη πως αυτό θα ικανοποιούσε όλους και η Ευρώπη θα είχε πολύ περισσότερες ε, επιτυχίες από ότι τώρα. Αυτά προς το παρόν. Παραμένω ε, ανοιχτή στα σχόλια και στις ερωτήσεις σας. Σε παρακαλώ περάστε από το γραφείο μου ή πάρτε με τηλέφωνο. Με τα χαράς να συζητήσω μαζί σας ό,τι θέλετε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Βίξτρομ. Να σας υπενθυμίσω ότι η προθεσμία για τις τροπολογίες είναι η 3η 10 Σεπτεμβρίου, 12 το μεσημέρι. 10 Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι λοιπόν. Αυτή είναι αναδιατύπωση, έτσι. Έχουμε μόνο τροπολογίες που αναφέρονται στην αναδιατύπωση της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μόνο αυτές. Τώρα λοιπόν είμαστε έτοιμοι για την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Έχουμε πολλά πράγματα να ψηφίσουμε. τέσσερι εκθέσει, τέσσερα θέματα και δεν φαίνεται πως θα έχουμε και δύσκολη ψηφοφορία. Θα είναι σχετικά απλά τα πράγματα, όπως και να έχει όμως. Ας αρχίσουμε. Γιατί έχουμε ώρα έχουμε θέματα. Σας παρακαλώ λοιπόν, προσέξτε να έχετε μαζί σας τις ε, ηλεκτρονικές σας κάρτες, να είστε έτοιμοι για την ψηφοφορία, για να γίνουν όλα πιο εύκολα. Κυρία Head, θα θέλετε να σχολιάσετε? Αν και η εκθεσή σας δεν, δεν είναι η πρώτη που ψηφίζουμε. Θα θέλατε να κάνετε κάποιο σχόλιο. Παρακαλώ. Ησυχία στην αίθουσα. Ετοιμαζόμαστε για την ψηφοφορία. Ναι, συγγνώμη, αλλά ξέχασα την ηλεκτρονική μου κάρτα στο σπίτι. Την ξεχάσατε, λοιπόν, λέει ο πρόεδρο. Ωραία. Γιατί δεν μπορείτε να ψηφίσετε με το χέρι. Αλλά παρακαλώ, όσοι από εσά δεν έχετε ξεχάσει τις ηλεκτρονικές σας κάρτες, να τις χρησιμοποιήσετε, να τις έχετε έτοιμες. Και Ας αρχίσουμε. Λοιπόν, από την αρχή θα τα πάρουμε. Καταρχάς η πρώτη ψηφοφορία αφορά την έκθεση της κυρίας Μαρίκια Γκάμπριελ για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων βραχίας διαμονής στους πολίτες της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακροτηρίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Τι έχουμε λοιπόν. 42 ψήφοι υπέρ, μία κατά, καμία αποχή. Αυτά ήταν. Τελειώσαμε. Σας ευχαριστώ κυρία Γκάμπριελ. Τώρα, πάλι έκθεση της κυρίας Γκάμπριελ για τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακροτηρίου για την επανεισδοχή προσώπων που διαμένουν χωρίς άδεια. Αρχίζουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 36 ψήφοι υπέρ, 7 ψήφοι κατά, καμία αποχή. Εγκρίνατε λοιπόν. Σας ευχαριστώ κύριε Κάπριελ, συγχαρητήρια. Έκθεση τώρα του κυρίου Ραούλ Ρομέβα για την εφαρμογή της οδηγίας του Συμβουλίου για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία. Έχουμε τώρα ορισμένε τροπολογίε να ψηφίσουμε. Ετοιμαστείτε. Αρχίζουμε. Τροπολογία 1. Υπέρ.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 κατά, αποχές, ε, απορρίπτεται. 12 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 13 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 14 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 15 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 16 υπέρ, ηλεκτρονικός έλεγχος, ηλεκτρονικός έλεγχος για την 15. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 21 ψήφοι υπέρ 22 κατά απορρίπτεται με μία ψήφο διαφορά. 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται και αυτή. 17 υπέρ κατά. Αποχές απορρίπτεται. 18 έχουμε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα έχει αποσυρθεί. Ψηφίσουμε το δεύτερο λοιπόν. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 20. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρολικός έλεγχος για την 21 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 22 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για το κείμενο όπως έχει τροποποιηθεί. Άρχεται η ψηφοφορία. Η 25 υπέρ 3 κατά. Ευχαριστούμε τον κύριο Ρωμέβα. Είχαμε 6 εποχές, ωστόσο... 16 εποχές, ωστόσο εγκρίθηκε. Τέταρτη ψηφοφορία για την έκθεση της κυρίας Χέντ για την τροποποίηση του κανονισμού σχετικά με τις πρόδρομες ουσίες ναρκωτικών. Άρχεται η ψηφοφορία. 39 ψήφοι υπέρ, 4 κατά, μία αποχή. Ευχαριστώ πολύ κυρία Χέντ. Αυτό ήταν. Δεν ήταν δύσκολο. Σας ευχαριστώ όλους. Προχωράμε τώρα στο σημείο 16. Οργανισμός για τη συνεργασία σχετικά με την επιβολή του νόμου και την κατάρτιση, Ευρωπόλ και κατάργηση των αποφάσεων 2009-371 του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Ο κύριος Αγκουστίν Τιαστεμέρα είναι ο εισηγητής. Είναι μια έκθεση προτεραιότητα η πρόταση τη Ευρωπόλη για την Επιτροπή μα. Θα ακούσουμε τον εισηγητή κ. Ντία Δεμέρα που θα μα παρουσιάσει το σχέδιο έκθεση και μετά τα υπόλοιπα μέλη που θα ήθελαν να παρέμβουν την ε, Επιτροπή και το Συμβούλιο Συμπεριλαμβανομένων. Θα ήθελα πριν ξεκινήσουμε να χαιρετήσω την παρουσία τη Κομισιόν και κάποιων καλεσμένων μας ε, ο κύριος Κάρλος Βάσκες από την ε, μόνιμη αντιπροσωπεία της Ισπανίας ε, αξιωματική Σύνδεση της Ευρωπόλ και μια ομάδα φοιτητών μαθητείας του δεύτερου έτους ε, από τη Σχολή Αστυνομίας Τσάβιλα. Καλώς ήρθατε. Ο κύριος Δία Δεμέρα. Muchas gracias, señor Presidente. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Και επαναλαμβάνω και εγώ το καλωσόρισμα προς τους Ισπανούς αστυνομικούς, τον, εκπρόσωπο της μόνιμης αντιπροσωπείας. Συγγνώμη κύριε Ντεμέρα, λέει ο πρόεδρος. Και εγώ ίδιος ξέχασα να αναφερθώ σε ένα ατύχημα το οποίο έλαβε χώρα στην Άβυλα, στην Ισπανία, ε, όπου έχασαν τη ζωή τους εννέα άτομα. Ε, εκφράζω ότι λείπουν και τα συλληπιτήριά μου ε, στους, ε, στους ανθρώπους που έχασαν τους δικούς τους σε αυτό το ατύχημα. Ήμουν και εγώ δήμαρχος της Άβυλα παλιότερα, οπότε με, πειράζει, με συγκινεί ιδιαίτερα. Ε, ο κ. Δεμέρα, κάνω και εγώ δικά μου τα λόγια σας, τα συλληπιτήριά σας προς τους ανθρώπους της Άβυλα. Ε, τι συνάλφη, Ε, νομίζω ότι έχουμε διανύσει ένα μεγάλο διάστημα που κορυφώνεται τώρα. Ε, η Ευρωπόλ χαρακτηρίζεται πρώτον από τη σήμαση του 1995, τα τρία πρωτόκολλα που, του 2007, την απόφαση του Συμβουλίου του 2009, για την οποία ήμουν επίσης ηγητής, και τέλος η κορύφωση, ο κανονισμός Ευρωπόλ, το, για τον οποίο συζητούμε σήμερα. Σύμφωνα με το άρθρο 88 της Συνθήκης Λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, λαμβάνουμε υπόψη, το οποίο λαμβάνουμε υπόψη λέγεται, λέει ότι το άρθρο το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο μέσω κανονισμού σύμφωνα με την ε, συνήθη ε, νομοθετική διαδικασία θα καθορίσουν τη λειτουργία, τη δομή, το πεδίο ε, λειτουργίας και τις αρμοδιότητες της Ευρωπόλη. Συνεπώς, κατόπιν της λήψης της ε, νομοθετικής πρότασης από πλευράς της ε, Κομισιόν, κάτι που έγινε σε 7 Μαΐου, ε, υπέβαλα 129 τροπολογίες στο νομοθετικό κείμενο την Κομισιόν. Κάτι που καταδεικνύει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι ε, αξιολογώ πολύ θετικά το νομοθετικό κείμενο και δεύτερον, ε, ότι πιστεύω πως πρέπει να βελτιωθεί. Οι τροπολογίες ε, ομαδοποιούνται σε τέσσερις κατηγορίες. Πρώτη κατηγορία ε, είναι η πιο περίπλοκη που αναφέρεται στην μη συγχώνευση Θεπόλ και Σεπόλ και Ευρωπόλ. Ε, δεν συμφωνώ με αυτή τη συγχώνευση. Οπότε ένα τμήμα των τροπολογιών ε, έχει ως στόχο την αποφυγή αυτής της συγχώνευσης. Δεύτερο, δεύτερη κατηγορία τροπολογιών έχει σχέση με κάτι που ενδυναμώνει, δίνει ζωή στην Ευρωπόλ και αναφέρομαι στον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Καμία αστυνομική υπηρεσία του δημοκρατικού κόσμου δεν μπορεί να ε, διαφεύγει του απαραίτητου κοινοβουλευτικού ελέγχου. Είναι απαραίτητος για να εξασφαλιστεί η διαφάνεια, για να εξασφαλιστεί η νομική ασφάλεια. Είναι απαραίτητος για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα της αστυνομικής δράσης. Ένα τμήμα των τροπολογιών μου έχουν ως ε, στόχο την εξασφάλιση αυτού του κοινοβουλευτικού ελέγχου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβουλία τρίτη κατηγορία τροπολογιών, τρίτη ομάδα, δέσμη τροπολογιών, ε, σχετίζεται με ένα ισχυρό σύστημα προστασίας των δεδομένων. Εδώ και πολύ καιρό λέω ότι στην βάση δεδομένων της Ευρωπόλ λείπει ακριβώς ένα σκέλος που είναι αυτό το σύστημα προστασίας των δεδομένων. Υπάρχει ένα τέτοιο σύστημα, αλλά θα πρέπει να βελτιωθεί ε, μέσω της βοήθειας του Ευρωπαίου ε, ε, επιπληκτηρητή. Τέταρτον, ε, θέλω να βελτιώσω την διακυβέρνηση της Ευρωπόλ. Είναι καλή ήδη. Και αυτό που προτείνει η Κομισιόν επίσης καλό, αλλά, θα, αλλά είναι λίγο χειρότερη από αυτήν που υπήρχε. Δεν συμφωνώ λοιπόν με την συγχώνευση σε Πολ ε, Ευρωπόλ. Οι περισσότερες πολιτικές ομάδες άλλωστε συμφωνούν μαζί μου. Ε, επίσης ε, συμφωνούν και οι γραπτές και προφορικές παρατηρήσεις ε, της Ευρωπολ και της ΕΠΟΛ, ε, οι γνώμες ε, των διευθυντών της ΕΠΟΛ και της Ευρωπόλ, όπως εκφράστηκαν εδώ στο Κοινοβούλιο, στην Επιτροπή Ελευθεριών, βρίσκονται στην κατεύθυνση που υποστηρίζω εγώ. Ακόμα και στο Συμβούλιο Τζάι 7 Ιουνίου 2013 τα περισσότερα κράτη-μέλη ήταν αντίθετα με την συγχώνευση. Γι' αυτό το λόγο ε, υποβάλλω τις συγκεκριμένες τροπολογίες. Μια ολόκληρη δέσμη. Ε, που έχει ως ε, στόχο του, την, την αποφυγή της σύγχρονης. Μετά, ε, ομάδα κοινοβουλευτικού ελέγχου που θα απαρτίζεται από τα Εθνικά Κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έτσι ώστε η, Ευρω... η Ευρωπόλ ε, να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις συνθήκης Λαβώνας. Ε, θα πρέπει οι δραστηριότητες της Ευρωπόλ να ελέγχονται από τους ερωτούς εκπροσώπους ε, των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο μηχανισμός ελέγχου των δραστηριοτήτων της Ευρωπόλ από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων προτείνω να γίνεται μέσω ενός μιας ομάδας κοινοβουλευτικού ελέγχου με μια μικρή ειδικευμένη δομή ε, την, οποία θα ε, την οποία θα δημιουργήσουμε εμείς, η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, ε, μαζί με την Επιτροπή Εσωτερικών Υποθέσεων των καθενός από τα Εθνικά Κοινοβούλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτός ο, αυτή η μονάδα αυτή η ομάδα θα έχει έδρα στο Ευρωπαϊκό ε, θα συγκαλείται από τον ε, πρόεδρο ε, της αντίστοιχης ομάδας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα συμπροεδρεύει εκπρόσωπος της Κομισιόν και ένας εκπρόσωπος και μάλλον και, και, και ένας εκπρόσωπος από την χώρα που θα έχει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτή την ομάδα ελέγχου, κοινοβουλευτικού ελέγχου, θα παρουσιάζεται και θα συζητείτε λέω θα παρουσιάζεται και θα συζητείτε έτσι το υπογραμμίζω αυτό η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της Ευρωπόλ το πρόγραμμα εργασίας ετήσιο και πολιετές η ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Μελτή ε, ε, Προστασίας ε, των Προσωπικών Στοιχείων και η έκθεση αξιολόγησης που, κάνει, που θα κάνει η Κομισιόν κάθε πέντε χρόνια για την αποτελεσματικότητα της Ευρωπόλ. Η, η ίδια ομάδα θα μπορεί να καλεί ε, τους υποψήφιους για εκτελεστικό γραμματέα της Ευρωπόλ ε, και για να ε, ενημερώνουν για τις, και για ενημερώνουν για τις δραστηριότητες του. Επίσης θα εμφανίζεται σε αυτή την ε, ομάδα ο εκτελεστικός ε, διευθυντής ε, της Ευρωπόλ, η υπηρεσία, Διευθυντής Υπηρεσίας Προστασίας Δεδομένων, η Κομισιόν και άλλοι. Η τα Εθνικά Κοινοβούλια θα λαμβάνουν πληροφορίες από την Ευρωπόλ για την αξιολόγηση των απειλών, για τις στρατηγικές ε, ε, αναλύσεις της, ε, που σχετίζονται με τους στόχους της Ευρωπόλ και τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων που έχει ζητήσει η Ευρωπόλ κάθε φορά. Όλα αυτά χωρίς να ξεχνάμε το εξής, ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει και ως δημοσιονομική αρχή να ε, επιτελέσει το καθήκον του. Πιο συγκεκριμένα ε, θα λαμβάνει τις ε, δημοσιονομικές προβλέψεις την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Ευρωπόλ και άλλες παρόμοιες εκθέσεις. Σε ό,τι αφορά την ε, ε, έδρα της ΕΠΟΛ, ε, να πω ότι η συνάντηση Τζάιτ e στις 7 Σεπτεμβρίου, τρεις χώρες ζήτησαν την, η Ουγγαρία συγκεκριμένα, η Ελλάδα και η Ιταλία ζήτησαν και η Ισπανία, τέσσερις λοιπόν, ζήτησαν την, έδρα της, νέα έδρα της ΕΠΟΛ. Ε, η δική μου προσωπική γνώμη είναι προφανώς υποκειμενική αλλά και αντικειμενική ταυτόχρονα. Γνωρίζετε ποια είναι η άποψή μου, οπότε δεν θα την επαναλάβω σε ό,τι αφορά την καινούργια έδρα της ΕΠΟΛ. Η ενίσχυση τώρα της, του συστήματος προστασία των δεδομένων. Για να ενισχυθεί αυτό το σύστημα, εξέτασα πολύ προσεκτικά τις ε, συστάσεις του κυρίου Πίτερ Χάστινγκ. Μεταξύ αυτών πιο σημαντικές, τις οποίες σκεφτετώ, είναι ε, η ενοποίηση των εθνικών αρχών, ε, των σημείων επαφής δηλαδή, ε, μεταξύ Ευρωπόλ και κρατών μελών. Η Ευρωπόλ μπορεί να έρχεται σε επαφή κατευθείαν με τις εθνικές αρχές, αλλά θα πρέπει καταρχήν να ενημερώνει τα σημεία επαφής. Το κράτος μέλος ε, το οποίο κατέχει τα δεδομένα ε, τα οποία δίνει στην Ευρωπόλ θα πρέπει να δώσει την ε, σύμφωνη γνώμη του προκειμένου αυτά να δοθούν σε τρίτες χώρες ή σε διεθνείς οργανισμούς. Αυτή η συνένεση δεν θα πρέπει μάλλον θα πρέπει να είναι ρητή. Για την καλύτερη λειτουργία της Ευρωπόλ της δίνουμε την δυνατότητα να επεξεργάζει στοιχεία που προέρχονται από ιδιωτικούς φορείς, ιδιωτικές πηγές. Υπό την προϋπόθεση ότι η, εθνική, η εφαρμοστή εθνική νομοθεσία ε, επιτρέπει την ε, ε, άμεση μεταβίβαση τέτοιων πληροφοριών σε αστυνομικέ αρχές. Σε κάθε περίπτωση η Ευρωπόλ θα αποστέλει σε εθνικές αρχές όλα αυτά τα στοιχεία σε ό,τι αφορά τη βελτίωση της διακυβέρνησης. Η νομοθετική πρόταση βελτιώνει την ε, διακυβέρνηση Ευρωπόλ ε, και τις ε, διαδικασίες, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το Διοικητικό Συμβούλιο και τον Εκτελεστικό Διευθυντή. Έχει αποδειχθεί η αποτελεσματικότητα ε, της Ευρωπόλ και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που αντιπροσωπεύουν τα κράτη-μέλη θα εξακολουθούν να είναι οι επικεφαλής των αστυνομικών αρχών του κάθε κράτους μέλους ή αυτά που ορίζονται από κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με την εμπειρία τους στην λυσή αστυνομικών ε, υπηρεσιών και την εμπειρία τους ε, στο θέμα της συνεργασίας μεταξύ αστυνομικών αρχών. Υπάρχει δυνατότητα οι εκπρόσωποι αυτοί ε, να διορίζουν ένα αντικαταστάτη ε, για, σε περίπτωση απουσία τους. Απουσίας τους. Ε, μεταξύ των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η, ε, η έγκριση του ετήσιου προγράμματος εργασίας, η έγκριση του πολιτούς προγράμματος, του προπολογισμού της Ευρωπόλ, της ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων της Ευρωπόλ και των δημοσιονομικών κανόνων που εφαρμόζονται θα, από ένα κατάλογο τουλάχιστον τριών ε, υποψηφίων που θα υποβάλει μια ε, ε, επιτροπή θα εκλέγεται ο εκτελεστικός διευθυντής. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με απλή πλειοψηφία με κάποιες εξαιρέσεις. Κάτι που θα δώσει καλύτερη αποτελεσματικότητα στο έργο της Ευρωπόλ. Προκειμένου να εγγυηθεί με την καλή, οδηγία, η καλή λειτουργία της Ευρωπόλ, ο εκτελεστικός διευθυντής είναι ο, ο, δι, ο κατά νόμο υπεύθυνος εκπρόσωπος της Ευρωπόλ. έχει τα εξή καθήκοντα. Ε, προετοιμασία των ε, δημοσιοκών εγγράφων, των ε, εγγράφων προγραμματισμού που υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο και για την εκτέλεση του ετήσιου και πολίτου προγράμματος δραστηριοτήτων της Ευρωπόλ. Αλλά και άλλα καθήκοντα στα οποία δεν θα αναφερθώ. Για να ετοιμάσω την πρότασή μου και προκειμένου να βελτιώσω τη διαφάνεια, έχω συναντηθεί ε, έχω διοργανώσει 20 συναντήσεις μεταξύ αυτών ε, με, τον, ε, με την Ένωση για Διακυβέρνηση της Ευρωπόλ ιδιαίτερα για τον, έλεγχο, τον κοινοβουλευτικό έλεγχο της Ευρωπόλ και θα συναντηθώ στο μέλλον με τους κοιοδησηγητές το 3 Σεπτεμβρίου διεύρυνση παράταση περίοδου για την υποβολή τροπολογίων μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου πάνω από 120 δηλαδή μέρες προκειμένου να υποβάλουν οι συνάδελφοι τι τροπολογίε του, 120 μέρες από όταν εγώ παρουσίασα τι τροπολογίες μου, θα λάβω υπόψη τι ε, τροπολογίε ε, στις 17 Οκτωβρίου. Στις 17 Οκτωβρίου και προβλέπω ψηφοφορία στην Επιτροπή 4-5 Νοεμβρίου. Να τελειώσω λέγοντας ότι είμαι στη διάθεση των συναδέλφων οποιαδήποτε στιγμή της μέρας, οποιαδήποτε μέρα της εβδομάδας. Θέλω να σας ευχαριστήσω, ιδιαίτερα εσάς που θα με βοηθήσετε πολύ, κύριε Χόλφερ. Και την κυρία Αλφάνο, την κυρία, τον κύριο Ταβάρες, Ρουί Ταβάρες και τον Τίμωθη Κίρκοπ, που δεν τον βλέπω. Τέλος, την κυρία Έρνστ, που ήταν πάντοτε πολύ κοντά και πολύ στενά συνδεδεμένη με την εξέταση του θέματος. Δεν θα ήθελα επίσης να ξεχνάσω, να ξεχάσω να αναφερθώ την Βικτόρια Νταμίτσι που εκπροσωπεί την Κομισιόν και δουλεύει εδώ και πολύ καιρό στα, σε θέματα Ευρωπόλ, ε, δουλεύει πραγματικά πολύ καλά. Αυτά, Πρόεδρε. Ευχαριστώ λοιπόν για την τοποθέτησή σα και για την παρουσίασή σα. Λοιπόν, και τώρα προτείνω να ακούσουμε πρώτα τα μέλη που έχουν ζητήσει το λόγο. του σκιώδεις πρώτα απ' όλα. Και μετά θα δώσουμε τη δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην Προεδρία να μιλήσουν. Η κυρία Ματιέ, καταρχά, έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή μας, τον κύριο Ντεμέρα. Έκανε σημαντική δουλειά όσον αφορά την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Ο κύριος Ντεμέρα είναι εμπειρογνώμων από αυτών των θεμάτων της Ευρωπόλ. Αλλά και ευρύτερα είναι ειδικό για τα θέματα της αστυνομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι ειδικό για τα θέματα της Ευρωπόλ προφανώς εργάζεται επί σειρά ετών επ' αυτών. Προφανώς είναι αναγνωρισμένος για τις γνώσεις του στην Επιτροπή μας, αλλά και εντός των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων γενικότερα, εντός του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Γκοστίν έκανε αξιοσημείωτη δουλειά. Αξιοσημείωτη η πρόταση που μας παρουσιάζει, αλλά ήταν αξιοσημείωτη και η παρουσίαση. Ευχαριστώ αγαπητέ Αυγουστίν. Ε, η πρότασή σου που είναι μπροστά μας Συνάδελφοι, η πρότασή του είναι πληρέστατη, παρουσιάζει καλύτερη διακυβέρνηση αυτού του μεγάλου οργανισμού, μεγάλου οργανισμού που υποστηρίζουμε στην Επιτροπή ε, Πολιτικών Ελευθεριών, διότι συνεργαζόμαστε με το Διευθυντή στενά, αλλά συνεργαζόμαστε εκτός Επιτροπής ΛΥΜΠΕ και στην Επιτροπή ΚΡΙΜ που έχουμε δημιουργήσει συνεργαζόμαστε. Επί σειρά μηνών στην Επιτροπή ΚΡΙΜ συνεργαστήκαμε με την Ευρωπόλ και δράτω με τις ευκαιρίες για να ευχαριστήσω το προσωπικό της Ευρωπόλ και τον διευθυντή της Ευρωπόλ. Αγαπητέ Ογκουστίν, η προτάση σου για την καλύτερη διακυβέρνηση του οργανισμού με εκτελεστικό διευθυντή εντελώς ανεξάρτητο στο έργο του και στην προετοιμασία του προπολογισμού, το σχεδιασμό των εγγράφων που υποβάλλονται προς απόφαση στο Διοικητικό Συμβούλιο είναι κάτι πολύ σημαντικό και το υπογραμμίζουμε. Είναι βασικό σημείο. Ο κοινοβουλευτικό έλεγχος που μας προτείνει είναι θεμελιώδες σημείο. Το αναφέραμε και σε διάφορες συζητήσει. Σημαντικότατο θέμα. Και για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων είναι κάτι καινοτόμο και σημαντικότατο Σημειώνουμε επίσης διεύρυνση αύξηση της προστασίας των δεδομένων με μεταφορά δεδομένων ε, ε, ρητή αδεία και όχι σαν κάτι που υπονοείται προς τρίτες χώρες. Αυτό είναι πολύ θεμελιώδες στην πρότασή σου, πάρα πολύ σημαντικό. Σημείωσα επίσης και το θεμελιώδες θέμα μας απασχολεί τους τελευταίους μήνες. Τη θέση σου όσον αφορά τη συγχώνευση σε Πολ Ευρωπόλ. Κάτι που προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχει σαφέστατη θέση, την οποία αναστερνίζομαι. Αρνούμεθα τη συγχώνευση Πολ και Ευρωπόλ. Είναι σαφές ότι όσον αφορά την Ευρωπόλ πρέπει να ξεκάθαρη αποστολή, αυτή που είχε πάντα, και δεν θα πρέπει την κατάρτιση να τη συνδέσουμε με αυτό. Όσο μας αφορά, θέλουμε να γίνεται κατάρτιση και θέλουμε να διονυστεί κατάρτιση αστυνομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό συγχώνευση Ευρωπόλ και Σεπόλ δεν μας εξασφαλίζει διόνυση της κατάρτισης αστυνομίας στην Ευρώπη. Και διαχωρισμός ε, ε, μεταξύ των δύο οργανισμών όπως έχει τώρα εξασφαλίζει τη διόνυση της κατάρτισης των αστυνομικών. Ευχαριστώ λοιπόν για την πρότασή σου. Θα την υποστηρίξουμε. Μπράβο. Μπράβο για αυτά που μας έδωσες και μας πρότεινε σήμερα το πρωί. Έβγε. Ευχαριστώ, δεν δουλεύει το μικρόφωνο. Ζώσεφ Βάιντεν Χόλτσα. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω θερμά τον ε, εισηγητή για αυτή την ε, παρουσίαση, την λεπτομερή παρουσίαση και για την ε, δουλειά και τη δραστηριότητά του μέχρι τώρα στο θέμα αυτό. Η δραστηριότητά του μέχρι τώρα μας δείχνει ότι έχει εξετάσει λεπτομερώς το θέμα, ότι το γνωρίζει βάθος το χρονοδιάγραμμα το βρίσκω βέβαια αρκετά φιλόδοξο. Θα το ψηφίσουμε ήδη στις 4 Νοεμβρίου. Αυτό το θεωρώ καλό. Όμως το πρόβλημα μου φαίνεται ότι αυτή η συγχώνευση Ευρωπόλ και Σεπόλ ενδεχομένως δημιουργήσει προβλήματα και χρειάζεται να πάρουμε ξεκάθαρες αποφάσεις, ότι υπάρχουν πάρα πολλά που πρέπει να ρυθμίσουμε. Το χρονοδιάγραμμα, επαναλαμβάνω, το θεωρώ πάρα πολύ φιλόδοξο. Όχι, όχι μόνο λόγω του περιεχομένου του, αλλά λόγω της σύνδεσης των δύο αυτών οργανισμών. Τώρα δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, αλλά να πω συνοπτικά ότι ο κοινοβουλευτικός έλεγχος και η βελτίωση που προτείνεται είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι μια πολύ σημαντική βάση για τις περαιτέρω εργασίες. Επίσης θεωρώ εξίσου σημαντικό να αναλάβει ο Ευρωπαϊκός ε, Εκπρόσωπος Προστασίας Δεδομένων ενεργό ρόλο. Πρέπει να πάρουμε στα σοβαρά την ε, κατάσταση αυτή. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ πολύ καλές και θετικές τις τροπολογίες σχετικά με, τον, με αυτό. Τώρα η βελτίωση της ε, δίκησης και η βελτίωση μέσω αυτής της ε, αποτελεσματικότητας ε, φυσικά είναι κάτι το οποίο θεωρώ θετικό. Τώρα, κάτι που μπορούμε να συζητήσουμε, διότι δεν με βρίσκει ακόμα απόλυτα σύμφωνο, είναι το γιατί θέλει να εξαιρέσει την, ε, το εκτελεστικό συμβούλιο εισηγητής. Πιστεύω πως χρειάζομαστε να το εξηγήσουμε αυτό, έτσι ώστε να καταλάβω και εγώ τι ακριβώς εννοεί. Πάντως, σε γενικές γραμμές θεωρώ πως αυτά που έχουν προταθεί θα οδηγήσουν σε πολύ θετικές εξελίξεις και ελπίζω να προλάβουμε να ολοκληρώσουμε το θέμα αυτό πριν το τέλος της νομοθετικής περίοδου. Το κύριο πρόβλημα όπως είπα, είναι το θέμα της ΕΣΕΠΟΛ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κέρκοπ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω καταρχάς ότι γνωρίζω πως σε αυτήν την Επιτροπή Ήμασταν πολύ τυχεροί επειδή η Europol μας ενημερώνει τακτικά για τις δραστηριότητε της. Είμαι σε στενή συνεργασία με τον διευθυντή της, τον κύριο Wainwright και πιστεύω πως ο ρόλος που παίζει η Europol σαφώς περιορίζεται από τον ορισμό των αρμοδιοτήτων της, όμως τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζουμε όλο ένα και μεγαλύτερες προκλήσεις ε, από πλευράς ε, αρχών επιβολής ενόμου, όπως της ε, Ευρωπόλ. Και πιστεύω, κύριε Πρόεδρε, ότι η συνεργασία των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος είναι κάτι πάρα πολύ βασικό και κάτι αποδεδειγμένο εξάλλου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς να δούμε ακριβώς το πώς μπορεί να γίνει πιο αποδοτική και αποτελεσματική Ευρωπόλ. Φυσικά ε, συμφωνώ απόλυτα με τα σχόλια του εισηγητή για τη συγχώνευση σε Πολ και Ευρωπόλ. Η ομάδα μου δεν θα υποστηρίζει κάτι τέτοιο. Ε, εντάξει, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας λέει ότι πρέπει να κάνουμε οικονομία, όμως δεν βλέπω πώς θα γίνει κάτι τέτοιο. Πιστεύω πως θα δημιουργηθεί μεγαλύτερη σύγχυση στους ρόλου και τις αρμοδιότητες των δύο αυτών οργανισμών. Δεν το υποστηρίζω λοιπόν. Ωστόσο, η πρόταση να διασφαλιστεί ένα ε, σαφή ε, μηχανισμός ανταλλαγής δεδομένων ανάμεσα στην Ευρωπόλη και τον ιδιωτικό τομέα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς, ιδιαίτερα σε σχέση με τα υπόλοιπα θέματα που ε, διαπραγματευόμαστε, που έχουν να κάνουν με προστασία δεδομένων. Επίσης, όσον αφορά την υποχρεωτική φύση της ε, ανταλλαγής πληροφοριών, πιστεύω πως ε, δεν χρειάζεται. Μια χαρά τα πήγαμε με την εθελοντική ανταλλαγή δεδομένων. Ορισμένες ε, φυσικά αστυνομικές αρχές ανταποκρίνονται καλύτερα, αλλά πιστεύω πως το πρόβλημα με την υποχρεωτική ανταλλαγή δεδομένων είναι ότι θα επικεντρωθούμε στην ποσότητα και όχι στην ποιότητα. Και πιστεύω πως ε, πολλές φορές είναι καλύτερα να έχουμε κάποιον προαιρετικό διακανονισμό παρά κάποιον υποχρεωτικό. Συνεισφορά τώρα στο αναλυτικό έργο της Ευρωπόλ. Παρατηρείται μια αύξηση του όγκου των ε, δεδομένων και της ε, κίνησης δεδομένων. Δεν ξέρω λοιπόν εάν αυτό καθιστά κάποια νομική υποχρέωση. Να σας πω ότι ο όρος νομική υποχρέωση με ανησυχεί. Δεν πιστεύω πως είναι απαραίτητο. Καλύτερα να υπάρχει μια προσέγγιση ω ιδίας πρωτοβουλίας. Τώρα, κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι εγώ προσωπικά θα ήμουν υπέρ του καταμερισμού κονδυλίων προς την Ευρωπόλ ανάλογα με τις αρμοδιότητες που θα αναλαμβάνει και σε σχέση με την συμφωνία SWIFT και με την συμφωνία για τα, την κατάσταση των επιβατών. Να σας πω ήδη ότι η συμφωνία SWIFT έχει ε, υπερφορτώσει τους υπαλλήλους της Ευρωπόλ από όγκο δουλειάς δεν ξέρω πώς μπορούμε να τους κάνουμε, να τους δώσουμε περισσότερη δουλειά. Φυσικά, επίσης να πω ότι είμαι υπέρ της, ε, του διεξοδικού ελέγχου, είμαι όμως και υπέρ της ε, αντελεγής πληροφοριών. Τώρα δεν είμαι σίγουρος εάν, αυτό, εάν η αλλαγή στο Διοικητικό, στο Εκτελεστικό Συμβούλιο και η περισσότερη ανάμειξη του Κοινοβουλίου στις εργασίες της Ευρωπόλη θα είναι κάτι που θα βοηθήσει και θα διευκολύνει τη λειτουργία της. Ωστόσο, καλωσορίζω τα σχόλια του εισηγητή, θα τον στηρίξω απόλυτα σε αυτά που θέλει να κάνει και πιστεύω πως το αποτέλεσμα θα είναι μια καλύτερη Ευρωπόλη, μια καλύτερα εξοπλισμένη Ευρωπόλη για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του 21ου αιώνα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριο Σταβάρες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον συνάδελφο Ντεμέρα, εξαιρετικό συνάδελφο και φίλο, να, τον, να σε ευχαριστήσω για αυτή την πολύ καλή δουλειά σου στο θέμα της Ευρωπόλη. Ε, η προσαρμογή συνθήκη της ε, Λισαβόνας ε, διαφόρων νομοθετικών κειμένων και ιδιαιτέρως του θέματος Ευρωπόλ θα πρέπει να είναι κάτι παραπάνω από ένα γραφειοκρατικό στάδιο. Θα πρέπει πραγματικά να ασκήσουμε πλήρως τις αρμοδιότητές μας. Και νομίζω ότι αυτό έκανες. Σε ό,τι αφορά τι τέσσερι δέσμες τροπολογιών για τις οποίες, ε, στις οποίες Καταρχήν το θέμα της συγχώνευσης της ε, αστυνομική Ακαδημίας με την Ευρωπόλ. Ε, το έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν. Γενικά οι κοινοβουλευτικές ομάδες υποστηρίζουν τη θέση σου. Πιστεύουμε ότι η αστυνομική κατάρτιση δεν θα πρέπει να συγχωνευτεί με την ε, ε, επεξεργασία στοιχείων. Ε, δεν είναι δυνατόν να δημιουργήσουμε ένα αμάλγαμα με τα Ευρωπόλ και Σεπόλ. Σε ό,τι αφορά την Σεπόλ και την έδρα της, υπάρχουν όπως είπες πολλές χώρες που ενδιαφέρονται. Τα κριτήριά μας όμως δεν θα πρέπει να είναι υποκειμενικά, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη αντικειμενικά κριτήρια. Αξιολογήσουν όπως αυτές τις ε, ε, ε υπηρεσίες ανθρωπινών δικαιωμάτων στις ε, υποψήφιες χώρες. Θα πρέπει δηλαδή ο καθεσμός της έδρας ε, να γίνει σύμφωνα με το κριτήριο της καλής συμπεριφοράς ό,τι αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα και την προστασία των δεδομένων στη χώρα η οποία θα λάβει την έδρα. Δεύτερη δέσμη, ε, κοινοβουλευτικός έλεγχος της Ευρωπόλ. Στις πρώτες μας συζητήσεις είχαμε πει ότι αποτελεί σημαντικό όρο προϋπόθεση για τη δική μας ομάδα. Η ε, Ευρωπαϊκή Ένωση αναλαμβάνει πλέον σιγά σιγά ε, υπερεθνικές αρμοδιότητες, συνεπώς αυτό θα πρέπει να συνοδεύεται από καλύτερο έλεγχο, κοινοβουλευτικό έλεγχο. Είναι ενδιαφέρουσα ιδέα δημιουργίας μιας ε, ιδιαίτερης ε, κοινοβουλευτικής ομάδας που θα παρακολουθεί το έργο της Ευρωπόλ. Περιλαμβάνεις και τα Εθνικά Κοινοβούλια εκεί. Ίσως αυτό θα μας δώσει τη δυνατότητα να διευρύνουμε τη συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Εθνικών Κοινοβουλίων. Ε, η συνεργασία αυτή μέχρι τώρα, παρόλο που συναντιόμαστε τακτικά, ίσως δεν έχει μια ενιαία μορφή, είναι κατακαιρματισμένη ως τώρα, δεν συγκεντρώνεται, δεν εστιάζεται, ίσως ε, αυτό είναι ένα καλό παράδειγμα για την βελτίωση αυτής της ανασίας στο μέλλον. Μία ερώτηση που θα ήθελα να σου κάνω είναι η εξής. Ε, τι γίνεται με την εγγύηση αυθεντικότητας των πληροφοριών που δίδονται. Η Ευρωπόλ λαμβάνει ε, στοιχεία μέσω ε, των ε, φάκελων των επιβατών, το PNR, μέσω του SWIFT κλπ. Έσω και, σε, και μέσω κλειστών συναντήσεων και μας δίδει στα κράτη-μέλη και σε εμά το Κοινοβούλιο δίνει τέτοιου είδους πληροφορίες. Καμιά φορά όμως δεν είναι ακριβής ή δεν είναι πλήρης, μπορεί να είναι και λαθασμένες Το πρόβλημα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και για τα κρατη και για τις τρίτες χώρες. Τέτοιου είδου περιπτώσεις ε, είναι προβληματικές. Και ενδεχομένως ε, ε τέτοιου είδου συμπεριφορές μπορεί να ε, είναι και αδίκημα. Πώς, μπορείς, πώς μπορούμε λοιπόν να βελτιώσουμε την, την εγγύηση ότι τα στοιχεία τα οποία δίνει η Ευρωπόλ ε, είναι αξιόπιστα. Αυτή η κοινοβουλευτική ομάδα ελέγχου, ε, όπως ε, είπες, μάλλον θα πρέπει να έχει ισχυρές αρμοδιότητες σε ό,τι αφορά και το διορισμό και την παράταση της θητείας ε, στελεχών της Ευρωπόλ. Ε, νομίζω ότι αυτό έχει άμεση σχέση με το προηγούμενο που είπα για την αξιοπιστία. Τέλος, για την προστασία των δεδομένων, συμφωνώ μαζί σου γενικά και θα υποβάλουμε, ε, θα υποβάλουμε σε αρκετές τροπολογίες για το εξής θέμα. Ε, πληροφορίες οι οποίες έχουν συλλεγεί με παράνομο τρόπο δεν θα πρέπει να μεταβιβάζονται. Αυτό έχει σχέση με το Prism αλλά και με το SWIFT, το, το, το PNR κλπ. Το Prism το ε, αφήσουμε εκτός διότι ε, δεν καλύπτεται από συμφωνίες με την, που έχει συνάψει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά οποιασδήποτε άλλες πληροφορίες συλλέγονται παράνομα δεν θα πρέπει να μεταδίδονται δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται. Αυτό αποτελεί κίνητρο και για τις υπηρεμιστικές υπηρεσίες των κρατών μελών και των ΗΠΑ ε, προκειμένου να σέβονται την ομιμότητα. Αυτά προς το παρόν. Ε, Είμαστε στην διάθεσή σου για διμερείς επαφές ως σκιώδης ηγητής. Εγώ και οι υπόλοιποι σκιώδης ηγητές φαντάζομαι. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ernst είναι η επόμενη. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή διότι πιστεύω πως έχει αναφερθεί στα κέρια σημεία, στα σημεία τα οποία μας ε, ενδιαφέρουν ε, περισσότερο. Πιστεύω πως ε, το θέμα αυτό είχε τον κατάλληλο εισηγητή, διότι δεν, ε, ήταν, ε, δεν είστε ιδεολόγος, αλλά πραγματιστής και πιστεύω πως αυτό το εκτιμούμε και ελπίζω πως θα καταφέρετε κιόλας να έχετε καλά αποτελέσματα. Τώρα, όσον αφορά την ΣΕΠΟΛ, την Αστυνομική Ακαδημία, σας στηρίζουμε. Πιστεύω πως η συγχώνευση δεν θα οδηγήσει σε εξοικονόμηση κονδυλίων αλλά σε σύγχυση. Πρέπει να δημιουργηθούν ε, νέες δομές, πρέπει να δοθούν νέα κονδύλια γι' αυτό, πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τον χώρο που θα συστεγαστούν αυτές οι δύο υπηρεσίες σε περίπτωση που θα συγχωνευτούν και πραγματικά δεν... Και πραγματικά να πω ότι η κατάρτιση στην αστυνομία είναι πιο σημαντική και, είναι και απαιτεί πολύ περισσότερες ε, δόμες από την Ευρωπόλη. Έχετε λοιπόν την απόλυτη στήριξή μας σε αυτό το θέμα. Δεύτερον, τώρα, ο κοινοβουλευτικό έλεγχο και η Επιτροπή Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, η επιτροπή αυτή που έχει προταθεί, μας βρίσκει σύμφωνους Και φυσικά θα μας απασχολήσει και εμάς η σύσταση αυτής της Επιτροπής Κοινοβουλευτικού Ελέγχου. Τι είναι όμως ο κοινοβουλευτικός έλεγχος. Ο κοινοβουλευτικός έλεγχος σημαίνει ότι στο ε, γραφείο μου θα έχω τα έγγραφα τα οποία χρειάζομαι. Δεν σημαίνει κοινοβουλευτικός έλεγχος ότι θα έρχεται η Ευρωπόλη εδώ και θα μας ε, ε, ενημερώνει γιατί τι γίνεται με το SWIFT και εμείς θα τους λέμε μπράβο, μπράβο, πολύ ωραία δουλειά σας. Όχι τελευταία φορά που ήρθε εδώ η Ευρωπόλ δεν ξέραμε τι γίνεται. Δεν θέλουμε λοιπόν μια, την πολιτική του μαύρου κουτιού. Θα πρέπει να το κάνουμε, αν θέλουμε να το κάνουμε σωστά, να το κάνουμε με τη σωστή μέθοδο. Και μπορώ να σας προτείνω λοιπόν τον τρόπο που, εργαζόμαστε, που εργάζονται αντίστοιχες επιτροπές κοινοβουλευτικού ελέγχου στη Γερμανία. Τώρα, τρίτο θέμα, προστασία δεδομένων. Αυτό το θέμα βρίσκει πολλούς να αιωρούνται πάνω από τα προσωπικά δεδομένα σαν του γήπε. Και αυτή τη στιγμή το βλέπουμε αυτό παντού, το βλέπουμε και στις διαπραγματεύσεις. Αλλά πρέπει να έχουμε υπόψη ε, πάντα ότι ένας, ε, αν θέλουμε να έχουμε έναν ε, σωστό κανονισμό για την Ευρωπόλη που να προστατεύει τα πνευματικά δικαιώματα νομικά, πρέπει να, λάβουμε, πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ τις νομοθετικές ρυθμίσεις που θα έχει αυτός ο κανονισμός. Τώρα, όσον αφορά την ε, αποτελεσματικότητα της διοίκησης και τις ενές δομές της διοίκησης. Πιστεύω πως εσείς ξέρετε καλύτερα από εμά πόσο αναγκαία είναι η αναδιάρθρωση και η εξυγίανση της ε, διοίκησης. Τώρα όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα αυτό ε, δεν μας βρίσκει και τόσο σύμφωνους, διότι αυτή η έκθεση είναι από τις σημαντικότερες εκθέσεις που έχουμε σε αυτή την νομοθετική περίοδο στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και μέχρι τα μέσα Σεπτέμβρη μας φαίνεται πως δεν μας φτάνει ο χρόνος, θα κάνουμε όμως ό,τι μπορούμε για να ε, καταθέσουμε τροπολογίες και να προχωρήσει το θέμα, αν και το βρίσκουμε ε, κάπως σε μικρό το περιθώριο. Αλλά πιστεύω ότι είναι πραγματικά αναγκαία να προχωρήσουμε και να κινηθούν τα νερά. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν πάρα πολλά καλά σχόλια. Στο τέλος θα έχετε δυνατότητα να δώσετε απαντήσεις. Η κυρία Κρίσμπεκ και μετά ο κύριος Κλάης και μετά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μετά το Συμβούλιο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα είμαι συντομότατη. Μιλούν ονόματι της Σόνια Αλφάνο που είναι άρρωστη και δεν μπόρεσε να είναι παρούσα σήμερα το πρωί. Προφανώς θα συμμετάσχει όμως σε αυτή την έναξη του διαλόγου που ο συνάδελφός μας ο Αγκουστίν ανακοίνωσε. Τις επόμενες εβδομάδες θα συμμετάσχει λοιπόν στην εμβάθυνση του διαλόγου το θέμα με τη σειρά μου και ονόματι της, και ομάδος να υπογραμμίσω το χαρακτήρα της ενδελεχούς αναλύσεως της εκθέσεως έξοχη δουλειά έγινε σαν βάση δουλειά που έκανε ο Αγκουστίν Δίας Τεμέρα και θέλω να πω όντας σύντομη ούσα σύντομη μάλλον, ότι η προστασία των δεδομένων είναι ένα θέμα που έχει γίνει ευαίσθητο. Σχετικά πρόσφατα. Είναι κάτι που ασχολεί τους πολίτες μας. Παρόλο που ήταν σήμα κατατεθέν της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, της δικής μας δεν θα υπενθυμίσουμε εμείς οι ίδιοι τους ε, ομοιρικούς διαλόγους που είχαμε για το SWIFT και για άλλα θέματα εδώ και κάποια χρόνια και η έκθεσή σας αγαπητέ συνάδελφε λαμβάνει υπόψη σωστά την ιδέα της ισορροπίας που πρέπει να εξευρεθεί μεταξύ προστασίας ελευθεριών από τη μια και της αναγκαίας καταστολής της εγκληματικότητας. Η ομάδα μας ακολουθεί την ίδια γραμμή. Όσον αφορά τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, δεν θα επανέλθω στα υποθέντα η ομάδα τα συμμερίζεται. Έχουμε ένα σημείο τριβής, πώς να το εκφράσω. Έχουμε ερωτηματικά, στο θέσουμε έτσι. Δεν θέλουμε να γίνει συγχώνευση σε πόλευρο Ευρωπόλ. Τις επόμενες εβδομάδες θα συνεχίσουμε την επεξεργασία του ζητήματος. Θέλουμε να βρούμε διεξόδους. Εντάχει λοιπόν Αυτή είναι η θέση της Σόνια Αλφάνο. Δράτω με τις ευκαιρίες που μου δίδεται για να ευχαριστήσω τους εκπροσώπους της Ισπανικής Αστυνομίας, πέραν αυτού όλες τις αστυνομικές δυνάμεις. Κυρίως ε, όσον αφορά τις, ε, τη διασυνοριακή προσέγγιση που ακολουθείται και ευχαριστώ τον Αγκουστίν για τη δουλειά που έκανε και την ανοιχτή του θέση. Ε, ε, ε, είναι ανοιχτό στο διάλογο και στην συγκεκριμένη ευρωπαϊκή οικοδόμηση. Είναι φημισμένος γι' αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κλέη έχει το λόγο. Σα ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα είμαι συντομότατος. Καταρχάς και εγώ θέλω να τονίσω ότι δεν έχω πιστεί απόλυτα κατά πόσο θα ήταν καλό να υπάρξει συγχώνευση σε Πολ και Ευρωπόλ και χαίρομαι που βλέπω ότι υπάρχει ε, αρκετή συνένεση από αυτού. Δεν πείθομαι εγώ με αυτή την ιδέα, ούτε ότι είναι επιχειρησιακά σωστή ιδέα. Ίσως θα είχαμε κάποιες οικονομίες. Μπορούμε να δώσουμε διάφορα παραδείγματα άλλα για την εξοικονόμηση χρημάτων. Αν δούμε ποιος είναι ο προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. υπάρχουν άλλοι τομεί που μπορούν να πραγματοποιηθούν οικονομίες και όχι εδώ. Είναι σημαντικό λοιπόν να παραμείνουν διαχωρισμένες οι δραστηριότητες της Ευρωπόλ από τις δραστηριότητες της ε, κατάρτισης. Έχω μία ερώτηση προς τον κύριο Δίας Δεμέρα. Θα ξέρετε ότι τώρα υπάρχει το θέμα συμφωνίας με τρίτες χώρες είναι ένα θέμα που τίθεται από πλευρά Ευρωπόλ για επιχειρησιακή συνεργασία με τις τρίτες χώρες. Επεξεργάζομαι μια σχετική έκθεση. Φαίνεται όμως να υπάρχουν πολλές επιφυλάξεις από πλευρά ομάδων, σκιωδών και νομικής υπηρεσίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δηλαδή ποια θα ήταν τα αποτελέσματα τέτοιων διαπραγματεύσεων. Ποιο θα ήταν το καθεστώς αυτών των διαπραγματεύσεων υπάρχει πρόταση για νέα οδηγία για την ίδια την Ευρωπόλ που έχει υποβληθεί. Ποια θα είναι η ισχύ των διαπραγματεύσεων και ενδεχομένων συμφωνιών που θα είναι αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων με τρίτες χώρες. Αν γίνονται διαπραγματεύσεις στα πλαίσια ενός συστήματος που θα αναδιαρθρωθεί μέσω νέας οδηγίας. Τίθενται πολλά ερωτηματικά όπως και για την προστασία των δεδομένων. Τελευταίο ερώτημα προς τον κύριο Ντίας Τεμέρα είναι το εξή. Η Ευρωπόλ θα πρέπει να ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις, να τις συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις ή θα πρέπει να περατωθούν πριν μπει στο νέο σύστημα η Ευρωπόλ. Πριν ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πάρει το λόγο, θα ήθελα να πω και εγώ κάποια πράγματα. Εκτιμούμε την πτυχή της προστασίας δεδομένων της εκθέσεως από τη συζήτηση σχημάτισα την εντύπωση ότι όπως και στην πρώτερη ακρόαση αυτή η ιδέα της συγχώνευσης σε Πολ και Ευρωπόλ δεν φαίνεται να πείθει πολλούς. Χαίρομαι που η μας αποφάσισε να αποσυρθεί η αναφορά στη συγχώνευση. Σαν επόμενο στάδιο χρειαζόμαστε ξεχωριστή πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη ΣΕΠΟΛ και ελπίζουμε αυτή η πρόταση να καταφτάσει σύντομα και να μπορέσουμε να επεξεργαστούμε το ζήτημα ξεχωριστά. Και να προχωρήσουμε και το θέμα της Ευρωπόλ. Η κυρία Αμίτσι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι παρούσα και θέλει να πάρει το λόγο, έτσι. Thank you very much, Madam Chair. Uh, firstly, I would like to... Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή κύριο Ντίας Δεμέρο, διότι έδωσε στις υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής τη δυνατότητα να συμμετέχουν στις πολλές συναντήσεις που έγιναν και με τους ασκιώδεις εισηγητές και με τα μέλη της Ευρωπόλ, έτσι ώστε να προετοιμάσει την έκθεσή του. Αυτό δεν ήταν μόνο χρήσιμο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ήταν και προνόμιο μας να είμαστε εκεί σε αυτές τις ε, συναντήσεις. Τώρα, θα ήθελα να κάνω μερικά σχόλια... για αυτά που συζητήθηκαν μέχρι τώρα, αρχίζοντας από τις ε, τέσσερις ε, δέσμες στην έκταση του κυρίου Διάς Δεμέρας. Τις τέσσερις δέσμες τροπολογιών, τις οποίες ανέφερα στην παρουσίασή του. και στις οποίες αναφέρθηκαν και άλλοι ευρωβουλευτές. Καταρχάς, όσον αφορά τη συγχώνευση, έχουν ήδη διεξαχθεί πολλές συζητήσεις για το θέμα αυτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει σημειώσει τις απόψεις που αναφέρθηκαν φυσικά και θα ήθελα εδώ να τονίσω ότι η Επίτροπος ε, Μάλιμστρομ έδωσε εξηγήσει ε, όσον αφορά ε, την πρόταση συγχώνευσης ε, σε Πολ και Ευρωπόλ την, στις 26 Φεβρουαρίου φέτος και μια δεύτερη φορά επευκαιρία της έγκρισης του νομοθετικού πακέτου στις 27 Μαρτίου. Ο εισηγητής σημείωσε ότι οι Υπουργοί δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων είχαν τη δυνατότητα να τοποθετηθούν για το θέμα αυτό στις 27 Ιουνίου. Έτσι λοιπόν δεν θα κάνω περαιτέρω σχόλια για αυτό. Τώρα, πώς γνωρίζετε, ο κοινοβουλευτικός έλεγχος και κυρίως η σύνδεση και ο σύνδεσμος των εθνικών κοινοβουλίων είναι κάτι που έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και βλέπουμε ότι και το Κοινοβούλιο έχει δώσει βάση σε αυτό και το θεωρούμε πολύ καλό. Το περιεχόμενο ε, της, ε, του ελέγχου αυτού ήταν ε, αυτό που απασχόλησε την Επιτροπή. Εμείς δεν θεωρήσαμε αναγκαίο να υπαγορεύσουμε λεπτομέρειες για τον, ε, για τον ε, διακοινοβουλευτικό συντονισμό του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Γι' αυτό λοιπόν η πρόταση του κυρίου Ντίας Δεμέιρα να συσταθεί μια επιτροπή κοινοβουλευτικού ελέγχου μας βρίσκει θετικούς όσον αφορά την προστασία των δεδομένων τώρα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέφερε ευθύ εξ αρχή, κατά την πρώτη παρουσίαση τη πρόταση αυτή, ότι η ενίσχυση τη προστασία δεδομένων ήταν ένα από του κύριου στόχου τη αναθεώρηση του νομικού πλαισίου τη Ευρωπόλ. Και ο κύριος Ντίας Δεμέρα θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικό το να υπάρχει η αρχή ιδιοκτησία σε των δεδομένων, δηλαδή τα κράτη-μέλη, οντότητα ή τα τρίτα μέρη που παρέχουν τα δεδομένα, να είναι εκείνοι που θα έχουν την κυριότητα των δεδομένων αυτών. Δηλαδή, θα πρέπει να δώσουν μια ρητή συγκατάθεση προτού μεταβιβαστούν τα δεδομένα αυτά οπουδήποτε αλλού. Επίσης, σημειώνουμε με μεγάλο ενδιαφέρον την πρόταση του κυρίου Δίας Δεμέρα για την δυνατότητα που θα μπορούσε να έχει η Ευρωπόλη να λαμβάνει δεδομένα από τρίτα μέρη. Αυτή η τροπολογία, από ό,τι καταλαβαίνουμε, έχει κατατεθεί για να ενισχύσει τις ε, δυνατότητες της Ευρωπόλη και να βελτιώσει την συλλογή πληροφοριών. Τώρα όσον αφορά την ε, διακυβέρνηση. Όπως ε, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εξηγήσει στο παρελθόν, η δομή της διακυβέρνησης που έχει προταθεί στον κανονισμό αντλεί πολλά στοιχεία από τα συμπεράσματα που εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή τον Ιούλιο του 2012 στα πλαίσια της κοινή προσέγγισης ε, ρύθμισης οργανισμών. Για παράδειγμα, η διαμόρφωση του Διοικητικού Συμβουλίου, τα καθήκοντα του Διευθυντή, η διαδικασία για τον ορισμό εκτελεστικού Διευθυντή, όλα αυτά ακολουθούν το μοντέλο που έχει δημιουργηθεί μέσω αυτής της οργανικής συνεργασίας που οδήγησε σε αυτή την κοινή προσέγγιση. Επίσης σε πολλές περιπτώσεις και οι λεπτομέρειες έχουν εμπνευστεί από τη λειτουργία άλλων οργανισμών. Επίσης, Σημείωσα ότι ο κύριος Εβάιντενχολτσερ μας ερώτησε για τον σκοπό της ε, συμπερίληψης ή μη ενός εκτελεστικού συμβουλίου. Να πω ότι ένα εκτελεστικό συμβούλιο θα ήταν ε, μια μικρή εκδοχή του Διοικητικού Συμβουλίου και αυτό το έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προαιρετικά. Δεν είναι υποχρεωτικό στοιχείο. Ο λόγος που το προτείναμε είναι ότι βασισμένη και πάλι και στις συστάσεις της κοινή προσέγγισης και στις κοινέ πρακτικές, έχει αποδειχθεί ότι μεγάλος όγκος δουλειάς που έχει σχέση με διοικητικά και οικονομικά ζητήματα του οργανισμού μπορούν να διαχειριστούν από αυτό, αυτή την μικρή, το μικρό συμβούλιο. Και έτσι λοιπόν το Διοικητικό Συμβούλιο θα μπορεί να επικεντρώσει την προσοχή του σε άλλα πιο βασικά ζητήματα. Επίσης, ο κύριος Κέρκχοπ αναφέρθηκε στην υποχρεωτική ανταλλαγή πληροφοριών. Και αν μου επιτρέψετε να τοποθετηθώ σε αυτό, θα ήθελα να πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι με την πρόταση κανονισμού καθίσταται σαφής η υποχρέωση που αναφέρεται στο εφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο και καθιστώντας την υποχρέωση λοιπόν αυτή σαφή, διευκολύνονται τα κρατημέλη ως προς την, ε, τον όγκο του, των δεδομένων που πρέπει να δώσουν στην Ευρωπόλ διότι αναφέρονται σαφώς οι τομείς ε, που πρέπει να δοθεί προσοχή και οι προτεραιότητες όσον αφορά τις εγκληματικές ενέργειες. Ε, ε, κύριο μέλημα λοιπόν με αυτή την πρόταση είναι να επικεντρωθούν τα κράτη-μέλη στους τομείς προτεραιότητας. Όχι να επικεντρωθούν στην συλλογή ενός μεγάλου όγκου δεδομένων μόνο και μόνο για να συμμορφώνονται με την υποχρέωση που θα έχουν. Ποιότητα τώρα ή ποσότητα. Θα ήθελα να σας πω εδώ ότι η Ευρωπόλ καταβάλει συνεχώς προσπάθειες για να παρέχει δείκτες στα κράτη-μέλη, δείκτες με τους οποίους θα μπορούν τα κράτη-μέλη μετά να βελτιώσουν την ποιότητα των δεδομένων. Αυτά προς το παρόν. Ελπίζω να μην μακρηγόρησα και θα χαρώ για τις επόμενες συζητήσεις. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, Ευχαριστώ να ζητήσω από την κυρία Πουλιακάιτε της ε, ε, Προεδρίας ε, αν θέλει να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχήν να ευχαριστήσουμε τον κύριο Ντίαθ για το έργο του. Περιμένουμε να συνεργαστούμε μαζί του για αυτό το θέμα. Πρόκειται για το πρώτο σημαντικό σημαντικό νομοθετικό κείμενο από τη Συνθήκη της Λισαβόνας που έχει σχέση με την ε, ε, εφαρμογή του νόμου, την επιβολή του νόμου. Το Συμβούλιο ε, διαφώνησε επίσημα στο Συμβούλιο Τζάι με την πρόταση Κομισιόν περί συγχώνευσης ΣΕΠΟΛ και Europol. Οπότε το κείμενο θα εξεταστεί χωρίς να γίνει λόγος για αυτό το ζήτημα. Η Προεδρία έχει προγραμματίσει μια σειρά ολοήμερων συνεδριάσεων της αντίστοιχης ομάδας εργασίας. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να εξετάσουμε την πρόταση, όχι μόνο σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, αν είναι απαραίτητο, θα τεθεί και σε υψηλότερο επίπεδο, προκειμένου το ζήτημα αυτό να προχωρήσει το συντομότερο δυνατό. Θα ήθελα λοιπόν να σας βεβαιώσω ότι και εμείς ε, επιθυμούμε μια ε, γρήγορη συνεργασία για την πρόθεση του θέματος. Ωραία. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Ο λόγος στον κύριο Ντίαθ Δεμέρα, τον εισηγητή. Ευχαριστώ, Κίνγκα. Ευχαριστώ όλους και όλους τους συναδέλφους ε, για τα σχόλιά τους. Ευχαριστώ Βερονίκ ως ε, εκπρόσωπο των, του ΕΛΚ για την καθαρότητα της σκέψης σου, για την υποστήριξή σου και για την ε, ε ρητή ε, απόρριψη της συγχώνευσης. Επίσης ευχαριστώ που συμφωνεί μαζί μου και για τις τρεις άλλες, το πνεύμα των τριών άλλων δεσμών. Ε, τροπολογιών. Σε ό,τι αφορά τον κύριο Όιντεν Χόλσερ, ε, ευχαριστώ καταρχήν για τα σχόλιά σου. Αληθεύει ότι είναι ανησυχητική η καθυστέρηση της ε, απόφασης για τη συγχώνευση. Αλλά εγώ είμαι ήσυχο γι' αυτό γιατί πηγαίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση. Η πλειοψηφία του Συμβουλίου και η πλειοψηφία του Κοινοβουλίου δεν επιθυμούν την συγχώνευση. Η κυρία Μάλστρομ επιμένει να μιλάει για συγχώνευση, αλλά νομίζω ότι θα καταφέρουμε να την πείσουμε. Το συντομότερο όμως θα πρέπει να μας υποπληθούν προτάσεις για τον κανονισμό ΣΕΠΟΛ και να τις εξετάσουμε. Κανονισμό ΣΕΠΟΛ συγκεκριμένα. Λέει ότι συμφωνείς με τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και με τη συναντήση με τον κύριο Χάστινγκ, τον επόπτη προστασία δεδομένων. Ε, για την ε, Τελεστική Επιτροπή έχω να πω το εξή. Το να κάνουμε μια φωτοτυπία του Διοικητικού Συμβουλίου ε, αλλά σε πιο στενή σύνθεση ε, τεσσάρων ατόμων θα έδινε υπερβολικά μεγάλη ε, εξουσία σε τέσσερα άτομα. Από την εμπειρία μου ε, προτιμώ να έχουμε πιο πλατιές δομές όπου θα αντιπροσωπεύονται όλα τα κράτη-μέλη. Όπως για παράδειγμα το Διοικητικό Συμβούλιο. Εξακολουθώ λοιπόν να έχω επιφυλάξει ό,τι αφορά την ε, Εκτελεστική Επιτροπή. Δεν λέω να υπάρχει κενό, γιατί ε, ο Γενικός ε, Γραμματέας εξακολουθεί να υπάρχει που και είναι το σημείο επαφής ανάμεσα στο ε, εκτελεστικό διευθυντή και το διοικητικό συμβούλιο. Για τον Τίμωθη, τον Τίμωθη Κίρκοπ. Ο Τίμωθη ήταν υπουργό εσωτερικών στο Ηνωμένο οπότε ξέρει πολύ καλά τη δουλειά αυτή. Ε, και εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ καλό το έργο της Ευρωπόλ και ο, ο διευθυντής ε, ήρθε, έχει έρθει επανειλημμένως εδώ να μας ενημερώσει για το ρόλο της Ευρωπόλ. Ε, και αυτός διαφωνεί με την συγχώνευση. Πολύ περισσότερο που οι Βρετανοί δεν θέλουν πλέον τη ΕΠΟΛ στο έδαφος τους. Σε ό,τι αφορά την υποχρεωτική ανταλλαγή πληροφοριών, το συνδέω με, τη, με τα όσα είπε η κυρία Νταβίτσι. Δεν είμαι υπέρ τη υποχρέωση. Η υποχρέωση την οποία αναφέρει τη Βικτόρια είναι μια έμεση, όχι άμεση υποχρέωση. Και άλλα Υπουργεία Εσωτερικών Κρατών Μελών μου είπαν ότι είναι πιο σημαντικό να εστιάσουμε στην ποιότητα παρά στην ποσότητα των δεδομένων. Υπάρχουν ε, δομές εσωτερικού ελέγχου στις οποίες δεν θα πρέπει το Κοινοβούλιο να παρέμβει και πρέπει να δώσουν περισσότερο περισσότερα χρήματα στην Ευρωπόλ, περισσότερε αρμοδιότητε σημαίνει μεγαλύτερη το προπολογισμό. Εσύ αναφέρθηκε στο SWIFT, ε, εγώ, ε, εγώ αναφέρομαι στο F3 για την καταπολέμηση του κυβερνοχώρου, του κυβερνοεγκλήματο, του εγκλήματο του κυβερνοχώρου. Ε, να, πρόσθετε αρμοδιότητε για τι οποίε χρειάζεται και πρόσθετη χρηματοδότηση. Για τον, ε, στον Ρουί Ταβάρης να πω ότι δεν είμαστε μόνο φίλοι, είμαστε κάτι πολύ παραπάνω από αυτό. Ε, Εκτός από τον ποταμό Ντουέρο ε, μοιραζόμαστε και άλλα πράγματα. Ε, η προσαρμογή στη συνθήκες της Αβωνάς των ε, ευρωπαϊκών οργανισμών είναι πολύ σωστό. Και πολύ περισσότερο που η Ευρωπόλ διαφέρει. Και εδώ θα διαφωνήσω με τη Βικτόρια. Ένα πράγμα είναι το, η συνολική εστίαση των ευρωπαϊκών οργανισμών και υπηρεσιών και άλλο η Ευρωπόλ. Και ο Ρουί Ταβαρές απορρίπτει την συγχώνευση. Ε, από, την άλλη φορά, από την άλλη μεριά για την έδρα της ΕΠΟΛ δεν έχουμε να πούμε πολλά πράγματα εμείς. Εγώ ε, μίλησα γι' αυτό. Πρώτον διότι είμαι πεπισμένος αντικειμενικά και δεύτερον διότι έχω τις δικές μου προσωπικές προτιμήσεις. Είναι και λίγο συναισθηματικό το ζήτημα. Ο, ο έλεγχος, έχει δίκιο ο Ρουί Ταβάρες, πρέπει να είναι ουσιαστικός. Και εδώ νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι, και η Κομισιόν και όλοι. Μέσω της ε, πρότασής μου πραγματικά ενισχύουμε τον ρόλο του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Ε, θα γίνεται μια τακτική τακτική συνάντηση, ο έλεγχος θα είναι τακτικός, ε, όχι ε, περιστασιακός. Ε, τελειώνω, Κίνγκα, αλλά πρέπει να απαντήσω σε όλους τους συναδέλφους για λόγους ευγένειας. Ε, Ρουί, ρώτησε. τι γίνεται με κάποιες πληροφορίες. Οι πληροφορίες έχουν τρεις διαβαθμίσεις αν, ανεξαρτήτως της ομάδας κοινοβουλευτικού ελέγχου υπάρχουν στα Εθνικά Κοινοβούλια και κοινοβουλευτικές ομάδες ελέγχου, πολύ περισμένη σύνθεση, ε, οι οποίες εξετάζουν διαβαθμισμένες πληροφορίες. Εκεί, σε αυτές τις επιτροπές, θα μπορούσε να ε, αναφέρει ε, ο διευθυντής της Ευρωπόλ, όπως επίσης και στην ομάδα κοινοβουλευτικού ελέγχου, σε πολύ περιορισμένο κύκλο και κεκλεισμένο των θυρών. Όλες οι πληροφορίες που δίδονται θα πρέπει να είναι νόμιμες, έχεις δίκιο, προφανώς νόμιμες. Κορνέλια. Κορνέλια, ευχαριστώ για τα λόγια σου. Και ευχαριστώ που διαφωνείς και εσύ με την συγχώνευση. Συμφωνείς με το κοινοβουλευτικό έλεγχο, θεωρείς θα πρέπει να είναι αποτελεσματικός και διαφανής. Ε, ζητάς να λάβουμε υπόψη την οδηγία που ισχύει αυτή τη στιγμή και να μην ξεχνάμε ότι ε, πρόκειται για μια αστυνομική δομή. Τώρα, για το χρονοδιάγραμμα κάποιες αμφιβολίες εκφράζει, θα το δούμε. Θα το δούμε. Κύριε Κρέσλε, ε, για την κυρία Αλφάνο παρακαλώ ε, μετάφερε της ε, τις ευχές μας για καλή ανάρρωση. Ε, ασφάλι θα πρέπει να ισορροπήσουμε ασφάλεια και ελευθερίες, πολύ σωστά. Ξέρω ότι στην ομάδα σας έχετε κάποιες επιφυλάξεις. Μ' ακούς? Όχι, δεν μ' ακούσε. Σου μιλάω. Ωραία, μα πού μ' ακούς. Ευγενέστατη. Ξέρω ότι στην ομάδα σας έχετε κάποιες επιφυλάξεις ό,τι αφορά τη σύγχυση, συγχώνευση. Ε, ωραία, καλό αυτό. Ελπίζω να εκφραστείτε εναντίον τη συγχώνευση. ο κύριο Κλά και αυτό κατά τη συγχώνευση. Και κάνει μια πολύ περίπλοκη ερώτηση. Είναι μια ερώτηση που έχει σχέση με τι συμφωνίε με τι τρίτε χώρε, αυτέ που ισχύουν ήδη και τι μελλοντικέ. υπάρχουν νομικά θέματα. Και έχουμε ζητήσει τη γνωμοδότηση τη νομική υπηρεσία όταν έχουμε την απάντησή τη. θα, σου αν θέλεις και Κίνγκα, πρόεδρος. Ευχαριστώ για τη θέση σου σε ό,τι αφορά τη συγχώνευση. Να σου διευκρινίσω το εξή. Μη με ευχαριστείς που ε, εγώ αφαίρεσα ε, από το κείμενο τις αναφορές για την συγχώνευση. Ξέρει η Βερονίκ ότι πάντοτε από παλιά ήμασταν εναντίον της συγχώνευσης για την Βικτόρια Νταμίτσι να την ευχαριστήσω και πάλι. Παρόλο που είναι πολύ νέα, πάντοτε μου μαθαίνει πράγματα. Ακόμα και όταν διαφωνώ, που διαφωνούμε συχνά, ε, βγαίνω πάντοτε σοφότερος. Ε, είναι αλήθεια ε, ότι η κυρία Μάλστρομ δύο φορές εξήγησε το σκεπτικό της και είναι αλήθεια ότι και το Σύμβουλιο έλαβε θέση. Ε, η Σεσίλια, η Βικτόρια σήμερα απλώς ε, σημειώνει σήμερα την, τη σημασία της ομάδας κοινοβουλευτικού ελέγχου και το θέμα της κυριότητας των δεδομένων. Ωραία, εντάξει, τα σημειώνει, θα τα σκεφτεί η Κομισιόν. Επίσης, σημείωσε και άλλα ζητήματα για την ποιότητα των δεδομένων κλπ. Ε, επίσης, σου είπα ήδη ότι η Ευρωπόλ δεν είναι ίδια με τις υπόλοιπες ε, υπηρεσίες και οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Και απάντησα και στην κυρία Ταβίνση σε ό,τι αφορά την ε, εκτελεστική επιτροπή. Ναι. Τελειώνω. Ευχαριστώ πολύ το Συμβούλιο για την παρέμβασή του. Ε, ευχόμαι καλή επιτυχία στη Λιθουανική Προεδρία. Και ε, ευχαριστούμε και για το πρόγραμμα των συνεδριάσεων που έχει καθορίσει. Ευχαριστώ πολύ για την έξοχη συζήτηση και την καλή δουλειά. 19 Σεπτεμβρίου είναι μια ημερομηνία που είναι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών και πρέπει να προχωρήσουμε τάχιστα διότι πήραμε είδηση ότι έχουμε άλλα δύο σημεία στην ημερήσια διάταξη πριν τις 12. Επόμενο, η κατάσταση μεριωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2012. Ο Μισέρ είναι συγητής που ετοίμασε δύο έγγραφα εργασίας και θα συζητήσουμε τα έγγραφα εργασίας και θα ακούσουμε την παρουσίαση του σχεδίου εκθέσεις της 30 ε, Σεπτεμβρίου Ζητώ από τον εισηγητή λοιπόν να συνοψίσει τα δύο έγγραφα εργασία και μετά θα δώσω το λόγο στα μέλη που θέλουν να συμβάλλουν στη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Κυρία Πρόεδρε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν σας μαθαίνω κάτι καινούριο εδώ, υιοθέτησε την περασμένη εβδομάδα την έκθεση του συναδέλφου Λουί Ταβάρες όσον αφορά την κατάσταση μελιωδών δικαιωμάτων στην Ουγγαρία συζητήθηκε η κατάσταση στη Βουλγαρία και πέρασαν ψήφισμα όσον αφορά την εποπτεία των Ευρωπαίων πολιτών από τι μυστικέ υπηρεσίε, την παρακολούθηση. Προφανώ είναι σαφέ τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι στο επίκεντρο των εργασιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, πήραν θέση όλο και πιο σημαντική στι δράσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όμω θα πρέπει να διαπιστώσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση περνά εδώ και αρκετού μήνε περίοδο κρίση. Η κρίση δεν είναι μόνο οικονομική, αλλά δυστυχώς και δημοκρατική. Η απόφαση της Ουγγρικής κυβερνήσεως ή η πρωτοβουλίε της Ρουμανικής κυβερνήσεως την περασμένη, το περασμένο καλοκαίρι κατά στη Βουλγαρία και η συστηματική παραβίαση κάποιων θεμελιωδών δικαιωμάτων σε κάποια κράτη-μέλη, όπως η Ιταλία στον αφορά τη δικαιοσύνη και την κατάσταση των φυλακών, παραδείγματος χάρη, όλα αυτά καταδεικνύουν σαφώς τις πολιτικές δυσκολίες που υπάρχουν και καμιά φορά και πρέπει να το παραδεχτούμε την έλλειψη πολιτικής βούλησης για την εφαρμογή των μηχανισμών που προβλέπουν οι συνθήκες καθώς και την ανάγκη να δημιουργηθεί ένας νέος μηχανισμός που θα εγκαιάται και θα ενισχύει το σεβασμό, την προστασία και την προώθηση των αξιών της Ενώσεως και αντιμετωπιστούν οι καταστάσεις κρίσεως στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε κάποια κράτη-μέλη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δημιουργήσει διάφορα όργανα για να εγγυηθεί το σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, τα κριτήρια τη Κοπενχάγη, τη συμπερίληψη των άνθρωπων 2 και 7 στη Συνθήκη τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω, τη Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, που στη Σύμβαση, Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. δυστυχώ, αυτό το κεκτημένο βασιζόταν σε μια υπόθεση που τελικά ήταν ανακριβή, Δηλαδή ότι η δημοκρατία και το κράτο δικαίου, τα θεμελιώδη δικαιώματα θα διατηρούνται και διαφυλάσσονται χωρί καμία ιδιαίτερη παρέμβαση τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Δυστυχώ αυτό απεδείχθη ανακριβέ από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όπως ανέφερα τα δικαιώματα του ανθρώπου πάντα ήταν και είναι στο επίκεντρο των δράσεών του. Υιοθετήσαμε κατά το παρελθόν σειρά εκθέσεων σε αφορά την κατάσταση των μελιωδών δικαιωμάτων και επίση ενδιαφερόμαστε πιο συγκεκριμένα σε κάποια δικαιώματα που απειλούνται όπω η ελευθερία των μέσων ενημέρωση και έχω υπόψη μου την Ιταλία και την Ουγγαρία εδώ, τα δικαιώματα των Ρωμά, Ιταλία, Γαλλία, τα δικαιώματα των ΛΟΑΔ, κυρίως Λιθουανία και Πολωνία, και εξετάσαμε και λεπτομερώς την κατάσταση εις Ουγγαρία. Στο πρόσφατο ψήφισμα για την κατάσταση μελωδών δικαιωμάτων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κυρίως υπογράμμισε την αναγκαιότητα επεξεργασίας μηχανισμών που θα εγγυώνται το σεβασμό, την προστασία και την πρόθεση των αξιών της Ενώσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη-μέλη. Υπάρχει ένα κενό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο θα πρέπει να ασκήσουν πιο ενεργό δράση όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα. Είναι ένα θέμα που τακτικά προωθείται, ένα επιχείρημα, είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει το δίλημα της Κοπενχάης όπως αποκαλείται ίτη. Αν οι υποψήφιες χώρες πρέπει να σέβονται τις δημοκρατικές αρχές, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα πριν προσχωρήσουν την Ένωση, δυστυχώς Κανένα αμέσω δεν προβλέπεται μετά την προσχώρησή τους, ώστε να επιβάλλει καιρό στα κράτη-μέλη που δεν σέβονται αυτές τις αρχές. Τούτου λεχθέντος η συνθήκη μας επιτρέπει ήδη τη δυνατότητα να ξεκινήσουμε εφαρμογή νέων μηχανισμών και νέων μέσων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πρωταρχικό ρόλο να παίξει στην, στην πρόταση νέων μέσων που θα έχουν στο στόχο την ενίσχυση σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στην Ένωση, δυνάμει της ισχυούσης συνθήκης και η αναγκαίων μέσω τροποποίησεων αυτής. Από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτή η αντιμετώπιση την παραβίαση των μελιών δικαιωμάτων προσφεύγοντα σε διάφορα μέσα όπω είναι διαδικασία κατά παράβαση, αναστολή προσωρινή των δεσμεύσεων των πρόωρων του Ταμείου συνοχή τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω, μηχανισμό συνεργασία και επαλήθευση, προειδοποίηση και πολιτικό διάλογο, τεχνικό διάλογο, συνεργασία με το Συμβούλιο τη Ευρώπη και άλλα δεσμικά όργανα και διεθνή όργανα. Και μετά με έδωσε προσανατολισμό όσον αφορά τη δικαιοσύνη ε, μόνο την, την, το αστικό δικαφορούσι και θα πρέπει μεσοπρόθεσμα να υπάρξει και άλλο μέσο που θα εφαρμοστεί. Αναφέρθηκε αναγκαιότητα τροποποίηση των συνθήκων, ανακοίνωσε ότι θα μπορούσε να προτείνει και σχέδια τροποποίηση των συνθήκων πριν το τέλο του 2013, αρχές 2014, για να οργανωθεί μια συζήτηση κατά διάρκεια των εκλογών συμπεριλαμβανομένου και το άρθρου 7 και ότι η συνένεση θα πρέπει να είναι εγγυημένη πριν να γίνει πρόταση. Η κυρία Ραντάιν ήδη ανακοίνωσε στην ε, Ολομέλη την περσμένη εβδομάδα ότι δρομολογείται μια ανακοίνωση επί του θέματο και ένα σεμινάριο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή επ' αυτού. Από πλευρά Συμβουλίου χαιρόμαστε ότι τα κράτη-μέλη συζητούν σήμερα τη δυνατότητα ενισχύσεω των ευρωπαϊκών μέσων που έχουν σαν στόχο τη διόρθωση των παραβιάσεων των αξιών τη Ενώσεω και ένα δημιουργηθεί νέο μηχανισμό που θα υποστηρίζει καλύτερη την προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων και την εφαρμογή του κράτου δικαίου στα κράτη-μέλη. Η παρούσα συνθήκη ήδη δίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση πολλέ αρμοδιότητε αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα, κυρίω μέσω των άρθρων 2 και 7, παράγραφο 1 τη συνθήκη όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμω αυτά τα άρθρα δεν ελήφθησαν υπόψη επαρκώ. Και ήγγει η ώρα να θεσπιστεί νέο μηχανισμό που θα εγγυάται το σεβασμό, την προστασία και την πρόθεση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των αξιών τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Επεξεργαζόμενοι δείκτε εξασφαλίζοντας την παρακολούθηση καταστάσεως εντός της ενώσεως, καθώς και εντός των κρατών μελών, προβαίνοντας κατά θέμα και κατά κάτω μέλος αξιολογήσεις, χρησιμοποιώντας τα σχετικά μέσα που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, αναπτύσσοντας και θεσπίζοντας διάφορες συστάσεις και κυρώσεις για την αντιμετώπιση των παραβιάσεων του άρθρου 2 της συνθήκης. Θέλω να είμαι σαφής. Μόνο ένας τέτοιος μηχανισμός μπορεί να εξασφαλίζει ότι όλα τα κράτη-μέλη με δίκαιο, ισότιμο, διαφανή και αντικειμενικό τρόπο θα εφαρμόζουν αυτές τις αρχές να μην υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά και διπλές προδιαγραφές θα πρέπει όλα τα κράτη-μέλη να αποδεχθούν να συμμετάσχουν στο μηχανισμό. Δυστυχώ, κάποιες χώρες στο Συμβούλιο ήδη κολλησιεργούν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορέσει να θετήσει απόφαση από αυτό των θεμάτων, κάτι που έκανε και την παρακολούθηση αναφορά τα θέματα τη διαφθορά Ευρωπαϊκή Ενώσεω και στα κράτη-μέλη και να προτείνει νέα μέτρα πολιτικής φύσεω εν συνεργασία με την ομάδα εμπειρογνωμών τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω, την Οργανισμό για τα Δικαιώματα και το Συμβούλιο της Ευρώπης. Το άρθρο 7 παράγραφο 1 δεν θα πρέπει να θεωρηθεί σαν μια πυρηνική βόμβα, αλλά σαν μια δυνατότητα να ξεκινήσει επίσημος και θεσμικός διάλογος μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και 100 μελών όταν υπάρχει ένας κίνδυνος παραβίασης σοβαρής των αξιών της ενώσεως. Επ' αυτού η ομάδα μου υπήρξε σαφέστατη. Το ότι δεν χρησιμοποιήθηκε μέχρι τώρα αυτό το μέσο και κυρίως όσον αφορά την Ουγγαρία οφείλεται, είναι προφανές, στην έλλειψη πολιτικής βούλησης και στο υψηλό επίπεδο ομοφωνής απαιτείται για να εφαρμοστεί. Συμφώνει ο γνώμης μας ακόμα και αν υπάρχουν κάποια σημαντικά θέματα που θα πρέπει ήδη να εξεταστούν και να επιληθούν στα πλαίσια της παρούσης συνθήκης, άλλα θέματα θα ίσως να χρειάζονται μια αναθεώρηση τη εν λόγω συνθήκης. Όμω η αναβολή δράσεων και αποφάσεων που θα μπορούσαν να θετηθούν για μεταγενέστερο προβληματισμό όσον αφορά την αναθεώρηση τη συνθήκη δεν αποτελεί ενδεδειγμένη απάντηση στι ανάγκε κατεπίγουσε όσον αφορά το σεβασμό και την προστασία και την πρόθεση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των αξιών των ιδρυτικών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Ήδη υπάρχουν πολλά μέτρα που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στο σεβασμό των αξιών που αναφέρονται στο άθρο 2 και θα μπορούσαν να εφαρμοστούν μέσως. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να επεξεργαστεί νέα μέσα ώστε να αντιμετωπιστεί η οικονομική κρίση και η χρηματοπιστική κρίση που αντιμετωπίζουμε τώρα. Θα έπρεπε τουλάχιστον να αποδείξει το ίδιο θάρρο και την ίδια αποφασιστικότητα στου τομεί που άπτονται των ελευθεριών, των δικαιωμάτων των Ευρωπαίων πολιτών και των αξιών από των οποίων εδράζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελπίζω ότι αυτά τα θέματα και οι προτάσεις που συμπεριλαμβάνονται στα δύο έγγραφα εργασία θα αποτελέσουν βάση για την ανάπτυξη, κατάρτιση της εκθέσεως για τα μερικά δικαιώματα και να υπάρξει επικοδημοτικός διάλογος μαζί σας καθώς και με τα άλλα θεσμικά όργανα στα πλαίσια μιας συζητήσεως δημοσίας που θα ξεκινήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά με του Συμβουλίου. Είναι θεμελιώδες να επιτρέψουμε επίσης και στους πολίτες να συμμετάσχουν σε αυτή τη συζήτηση και η προτεραιότητα είναι να μπει στο επίκεντρο τη έκθεση ο πολίτη, τα δικαιώματα και ελευθερίε. Αυτό έκανα. Το σχέδιο εκθέσεω θα υποβληθεί στην Επιτροπή τέλο Σεπτεμβρίου. Μέχρι τότε θα συναντηθώ με του κοιόδη συγητέ για να ανταλλάσσουμε απόψει και προτάσει, ούτω ώστε να επεξεργαστούμε σωστά την έκθεση. Επίση, προβλέπεται να οργανωθεί μια δημόσια κρόαση με τα άλλα θεσμικά όργανα, μη κυβερνητικέ οργανώσει, εμπειρογνώμονε και του πολίτε. Ευχαριστώ που με ακούσατε με θρησκευτική ευλάβεια. Ευχαριστώ πολύ για τα έγγραφα εργασία και για την παρουσίαση αυτή. Βλέπω ότι υπάρχει σύγκληση μεταξύ συμπερασμάτων Συμβουλίου, εκθέσεως, εκθέσεως ταβάρες της περασμένης εβδομάδας και των προτάσεων. Θα παρουσιαστεί το σχέδιο εκθέσεως στις 30 Σεπτεμβρίου. Τώρα έχουμε πολύ λίγο χρόνο στη διάθεσή μας. Ζητώ από όλους, λοιπόν, να μιλήσουν μόνο για ένα λεπτό ο καθένας για να δώσουμε κάποιες αντιδράσεις στον εισηγητή και μετά θα πρέπει να ολοκληρωθεί το σημείο της ημέρης διάταξης γιατί έχουμε κοινή συνεδρίαση στις 12 με την ΑΦΚΟ και τη Γιούρη νομίζω και, μετά πρέπει, και πρέπει να προετοιμαστούμε όπως καταλαβαίνετε. Η κυρία Μπάουερ είναι η πρώτη που θα πάρει το λόγο. Έχει το λόγο. Και παρακαλώ να είστε σύντομοι. Ευχαριστώ πολύ. Είναι λίγο δύσκολο να περιοριστώ σε ένα λεπτό για να πω όλα αυτά που θέλω. Έχω πάρα πολλά ερωτήματα για αυτή την έκθεση. Στην έκθεση αυτή μιλάμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά πραγματικά μας εκπλήσει το γεγονός ότι το περιεχόμενο δεν συμφωνεί με τον τίτλο, με τα θεμελιώδη δηλαδή δικαιώματα και την κατάσταση με τα θεμελιώδη δικαιώματα στην Ευρώπη. Δεν καταλαβαίνω τα άρθρα 2 και 3 της συνθήκης, τι σχέση έχουν με την έκθεση αυτή, σύμφωνα με τα άθρα αυτά, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει αρμοδιότητα να αποφασίσει, όχι το Κοινοβούλιο. Το Κοινοβούλιο δεν έχει αρμοδιότητα για αυτό το θέμα και πιστεύω πως ε, δεν μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα χωρίς αλλαγή των συνθήκων. Επίσης, από την έκθεση αυτή προκύπτει ένα άλλο ερώτημα. Τι γίνεται με, τα, με τη Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στην Ευρώπη. Διότι αυτό μπορούμε να το δούμε μόνο σε συνδυασμό με τα δικαιώματα στην Ευρώπη. Είναι νομικής φύσεως το ερώτημα. Και αυτό το νομικό ερώτημα είναι πολύ δύσκολο να το απαντήσουμε βασισμένοι σε αυτή την έκθεση. Πιστεύω πως πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στις ε, περαιτέρω διαπραγματεύσεις, διότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορεί να αντικαταστήσει το δικαστήριο. Τι θα κάνουμε με τις ε, δικαστικές αποφάσεις, ερωτώ. Τι γίνεται με τις ε, διαδικασίες επί παραβάση. Επαναλαμβάνω, το πρόβλημα αυτό δεν μπορεί να λυθεί χωρίς αλλαγή των συνθήκων. Για τον λόγο αυτό πιστεύω ότι αυτό το περιεχόμενο δεν είναι το κατάλληλο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Μπάουερ. Κυρία Στανόκα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Σημεριζόμαστε απόλυτα όλα όσα παρουσίασε ο κύριος Μισελ σήμερα στο κείμενο. Είναι μικρό το κείμενο, αλλά περιεκτικότατο και είναι μια καλή βάση για περαιτέρω συζητήσεις και ανταλλαγές απόψεων. Τώρα, θα ήθελα χάρη συντομίας να αναφέρω μόνο ότι η ομάδα μας έχει θίξει αυτά τα ερωτήματα και έχει επιστήσει την προσοχή στα προβλήματα εδώ και πάρα πολύ καιρό στα πλαίσια της ετήσιας έκθεσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Διότι οι εκθέσεις αυτές γίνονται ανακράτους Συνήθως αλλά στην περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει παρατηρηθεί ότι χρησιμοποιούμε διπλά στάνταρ και αρνιούμαστε να εξετάσουμε την κατάσταση σε ορισμένα κράτη-μέλη. Αρνούμαστε επίμονα, ιδιαίτερα όσον αφορά την ισότητα. Και βλέπουμε ότι, σε, ότι οι προτάσεις αυτές ε, κόλλανε στην εφαρμογή. Υπάρχει πρόβλημα δεν υπάρχει ενιαίος μηχανισμός ε, ταυτοποίησης για να επαληθεύσει το πώς ε, δρά ένα κράτος εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης υπάρχουν πάρα πολλές ε, ανησυχίες που προκύπτουν. Για παράδειγμα από την έκθεση Πέρνες. Για τη δική μου χώρα, τη Λετωνία, υπήρχαν πάρα πολλές ανησυχίες όσον αφορά το τι γίνεται με τα δικαιώματα των μειονοτήτων, με τους ανθρώπους ε, χωρίς ε, υπηκότητα, τους απάτριδες, με τα δικαιώματα των πολιτών ε, να συμμετέχουν σε τοπικές εκλογές. Όλα αυτά τα ζητήματα παραμένουν άλυτα. Δεν υπάρχουν τέτοια δικαιώματα δέκα χρόνια μετά από την έγκριση της έκθεσης και το πρόβλημα παραμένει. και ο λόγος που το πρόβλημα παραμένει είναι πολιτική αντίσταση από ορισμένε ομάδες. Στηρίζω απόλυτα την βελτίωση του μηχανισμού παρακολούθησης σε περιπτώσεις παραβίασης ανθρωπινών ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων. Επίσης έχουμε τον κύριο Κέρουμ εδώ, όπως και χθες. Και χθες ε, ήδη αναφέρθηκα σε αυτό το πρόβλημα που αναφέρθηκε και ο κύριος Μισελ, ότι ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων δεν έχει επαρκείς αρμοδιότητες για να ασχοληθεί με το θέμα αυτό. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δούμε πώς μπορούμε να δράσουμε στα πλαίσια των συνθήκων. Ευχαριστώ. Κύριε Βερζιά, έχετε το λόγο. Euh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ακούοντας τον Λουί Μισελ ε, με καθυσίχασε λίγο. Νομίζω ότι η έκθεση αφορά πραγματικά τα θεμελιώδη δικαιώματα και το θεσμικό κομμάτι μπορεί να γίνει αντιληπτό μόνο αν κάνουμε μια προηγουμένη ανάλυση της κατάστασης των θεμελιών δικαιωμάτων. Οι πολίτες ε, περιμένουν από μας να εντοπίσουμε τα προβλήματα ε, που υφίστανται σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ίσως αυτό θα μπορούσε να απαντήσει και στις, ε, εν μέρη στις ε, ε, επιφυλάξεις του ΕΛΚ. Αν και φοβάμαι δεν φτάνει. Μια ανάλυση της κατάστασης και, μια, και υπάρχει ένα θεσμικό κομμάτι. Ε, συμφωνώ λοιπόν με τις γενικές γραμμές της έκθεσης. βρίσκεται στο ίδιο μικρό σχήματος με την έκθεση Ταβάρες. Έχω όμως και κάποιες παρατηρήσεις να κάνω. Ένα από τα βασικά προβλήματα που θίγουν τα διεθνή όργανα και κυρίως Συμβούλιο της Ευρώπης και τα Ηνωμένα Έθνη, κύριε Μισελ, είστε εδώ. Αλλιώς να τα πούμε διμέρως. Ένα από τα βασικά προβλήματα λοιπόν που φύγουν τα διεθνή όργανα είναι το θέμα των μεταναστών εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως ούτε στο εγγραφό σας ούτε στις εισαγωγικές παρατηρήσεις νομίζω μιλήσατε για αυτό το ζήτημα. Και όμως είναι επικαιρό γιατί αφορά θέμα παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σχετικό με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η χάρτα των θεμελιών δικαιωμάτων εφαρμόζεται γενικά σε όλους όσους διαμένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο στους Ευρωπαίους πολίτες. Και μία άλλη παρατήρηση. Θεωρώ το ότι το άρθρο 7 είναι ε, ατομικό όπλο, πυρηνικό όπλο και δεν χρειάζεται, δεν χρειαζόμαστε καινούρια ε, νομικά εργαλεία. Αν εφαρμόσουμε το άρθρο 7 που δεν το εφαρμόζουμε, δεν θα αναφερθώ περαιτέρω σε αυτό το ζήτημα. Ορισμένοι συναλφοί και οι, Κομισιόν κρύβονται μονίμως πίσω από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το έχω βαρεθεί πια. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι πολιτικό όργανο που πρέπει να υποβάλει προτάσεις και πρέπει να καταγγέλει και κάποια πραγματάκια. ας μην στερούμαστε αυτή μας, αυτής μας δυνατότητας. Δεν το κάνουμε στα οικονομικά θέματα, ας, το, ας μην το κάνουμε ούτε και στα ανθρωπιστικά θέματα, θέματα δικαιωμάτων. Οι ευρωπαϊκές αρχές καλές είναι στη θεωρία, αλλά ακόμα καλύτερες όταν τις εφαρμόζουμε στην πράξη. Η αρχή κρατών κυβερνήσεων λοιπόν καλό θα ήταν να τις λαμβάνουν υπόψη τους στις, στην πράξη, στην πρακτική τους. Να μην μένουν μόνο λόγια αυτές οι ευρωπαϊκές αρχές. ξέρουμε ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά σε ό,τι αφορά το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην επικράτεια χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, Σε ό,τι αφορά τον Οργανισμό Θεμελιών Δικαιωμάτων, ε, καλόν είναι, ε, δεν έχουμε καταφέρει να του βοηθήσουμε πολύ. Ε, πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να του συμπερασταθούμε Η υπηρεσία αυτή δεν είναι πολιτική φύση. Εμείς είμαστε το πολιτικό όργανο, εμείς θα βγάζουμε τα συμπεράσματα από ε, τις πληροφορίες που μα δίνει η υπηρεσία θεμελιών δικαιωμάτων, ο Οργανισμό Θεμελιών Δικαιωμάτων. Ευχαριστώ. Κυρία Κίνκα Γκόντς. Ευχαριστώ πολύ. Όπως είπα και πριν, βλέπω μια μεγάλη σύγκληση ανάμεσα στις, στα, στα του Συμβουλίου, τα επιστολές των Υπουργών, την έκθεση, τα βάρες και το δικό σας έγγραφο εργασία τώρα. Και πιστεύω πως είναι καιρός να προχωρήσουμε. Βλέπουμε ξεκάθαρα πως έχουν τα πράγματα. Μιλάτε για δημοκρατική κρίση και όχι μόνο οικονομική κρίση στην Ευρώπη και πιστεύω ότι πραγματικά έχει έρθει η ώρα να προχωρήσουμε. Είναι και αυτός ο τρόπος να αποφύγουμε τα διπλά στάνταρ όπως έχει ήδη αναφερθεί πολλές φορές στην αίθουσα αυτή, να δημιουργήσουμε δείκτες, να διευρύνουμε το πεδίο εφαρμογή ε, του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων που ο οποίος πιστεύω πως είναι αρκετά έτοιμος να δημιουργήσει και να αναπτύξει αυτούς τους δείκτες. Και για εμάς θα είναι πολύ σημαντικό αυτό στο μέλλον να δούμε μια ξεκάθαρη εικόνα του τι γίνεται στην Ευρώπη, πώς τα διάφορα κράτη-μέλη αντιμετωπίζουν το κρατός δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα, το θεμέλιο δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό λοιπόν με τα χαράς να στηρίξω την πρότασή σας και ελπίζω το σχέδιο πρόταση ε, να, έχει, να είναι στα χέρια μας μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου. Κύριε Ταβάρης. Ε, Θα μιλήσω στα γαλλικά, μια και ο εισηγητής μας είναι γαλλόφωνος. Χαίρομαι που βλέπω ότι αυτή η έκθεση συνάδει με άλλες δουλειές που έχουμε κάνει στο παρελθόν εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δύο-τρία πράγματα έχω λοιπόν, να προσθέσω μόνο. Αυτή τη στιγμή όταν έχουμε στα χέρια μας την έκθεση θα έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε και περισσότερα σχόλια. Σε ό,τι αφορά τους δείκτες καταρχήν. Οι δείκτες είναι πολύ σημαντικοί και ιδιαίτερα όταν θέλουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση των θεμελιών δικαιωμάτων και της δημοκρατίας της χώρας μας. Δηλαδή, οι δείκτες είναι χρήσιμοι υπό την προϋπόθεση ότι η συνεργασία χαρακτηρίζεται από ε, αφοσίωση, ειλικρίνεια και προθυμία. Γιατί αλλιώς μπορώ να φανταστώ πώς θα λειτουργούσαν οι δείκτες. Με ανησυχεί το γεγονό ότι μπορεί να έχουμε ένα πολύ ωραίο πίνακα με δείκτε κλπ. Αλλά στην πραγματικότητα να υφίστανται σημαντικά προβλήματα τύπου του άρθρου 2. Παρόλο που οι δείκτες μπορεί να είναι εξαιρετικοί, λέω. Γι' αυτό και στην έκθεσή μου ψηφίστηκε την περασμένη εβδομάδα είχαμε προτείνει να ε, υπάρχει ένα σύστημα επιβεβαίωσης με την Επιτροπή της Κοπεχάγης. Έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι για την πραγματικότητα, θεσμική πραγματικότητα των κρατών μελών. Απ' την άλλη μεριά, άρθρο 7 Άρθρο 7.1 ξέρουμε ότι είναι ένα κέλυφος. Το 7.2 μπορεί να είναι πυρηνικό όπλο, αλλά ατομική βόμβα, αλλά ε, ε, από το 7.1 στο 7.2 η απόσταση είναι τεράστια. Και μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και πολλά διαδικαστικά εμπόδια. Είναι αλήθεια ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Τα κράτη-μέλη συνεργάζονται μόνιμα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη συζήτηση για την Europol διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν κρατημέλη που θέλουν να φιλοξενήσουν τη ΣΕΠΟΛ. Θα πρέπει τα κριτήρια του άρθρου 2 να ενταχθούν στις ε, πολιτικές αποφάσεις για τέτοιου είδους συνεργασία. Δηλαδή, αν δεν υπάρχουν εγγυήσεις ε, για την, τον διαχωρισμό των εξουσιών, ε, για την ακαιρεότητα της δικαιοσύνης, για την ακαιρεότητα και την ε, αμεροληψία των αστυνομικών αρχών κλπ. Τότε, αν υπάρχουν δηλαδή προβλήματα τύπου του άρθρου 2, δεν είναι δυνατόν να φιλοξενηθεί η έδρα και διάφορα άλλα τέτοια θέματα στα οποία θα μπορούσαμε να λάβουμε υπόψη την κατάσταση. Ευχαριστώ. Και τώρα ο κ. Λεμισέλο, εισηγητή, έχετε το λόγο για να ολοκληρώσουμε το θέμα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καταρχά, χαίρομαι που βλέπω ότι οι περισσότεροι που πήραν το λόγο, με την εξαίρεση τη κυρία Φορέλη, ε, θα προσθέσω την πίσω εκείνη, οι περισσότεροι συμφωνούν αρκετά με τι βασικέ γραμμέ του εγγράφου, των εγγράφων, των εγγράφων εργασία Μόνο έγγραφα εργασία είναι. Θέλουν να εμπνεύσουν. Μία διεύρυνση τη συζητήσεω. Να πω, κυρία Μπάουερ, ο εισηγητή θα υποστήριζε μία συζήτηση για τα θέματα που αναφέρεται στο δύο πρόγραμμα έγγραφα εργασία για να γίνει πιο θεσμική προσέγγιση στον την στα θεμελιώδη δικαιώματα και να γίνει δημόσια συζήτηση. Το ανέφερα. Θέλω συζήτηση. Να πω ότι πιστεύω ένθερμα όπως και η κυρία Σβερζιά, ότι είμαστε ένα κοινοβούλιο. Και σαν βουλευτές δεν μπορούμε εμείς να θέτουμε όρια στη σκέψη μας, ούτε στις πεπιθήσεις μας τις διντολογικές, ούτε ιδεολογικές ή πολιτικές. Ασκούμε πολιτική. Κανένας θεσμικός κανόνας δεν μπορεί να μας εμποδίζει να εκφράζουμε μία θέση και να εκφράζουμε προφανώς συστάσεις. Έτσι εξελίσσονται οι νομοθεσίε. Έτσι γίνεται και πραγματοποιείται η ανθρώπινη πρόοδο με την πάρα του χρόνου. Αλλά θα το συζητήσουμε. Κυρία Βερζά, βεβαίω στην έκθεση θα καλύψουμε σειρά θεμάτων που δυστυχώ δεν μπορέσαμε να συμπεριλάβουμε. Κλασική ελευθερίε, Κλασικές ελευθερίες, ελευθερία της έκφρασης, μέσα ενημέρωσης, δικαιώματα μειονοτήτων, ισότητα, μη διάκριση, μετανάστες, άσυλο, δικαιώματα παιδιών, ηλικιωμένων κλπ. Προφανώς θα έχουμε τη δυνατότητα να εμπλουτίσουμε το έγγραφο. Δεν σας κρύβω και θα δούμε πώς εξελιχθούν τα πράγματα και δεν απειλεί. Λοιπόν, προσωπικά πρέπει να σας πω ότι σχηματίζω ένα πίνακα στο μυαλό μου θεματικό με δείκτες και με χώρες. Ξέρω ότι δεν θα δεχτούμε βέβαια να κατονομάσουμε κάθε χώρα, αλλά ονειρεύομαι τέτοιο πίνακα. Δεν αποκλείω λοιπόν προσωπικά να συντάξω ένα τέτοιο πίνακα. Θα δούμε θα μπει σε παράρτημα ή όχι, αλλά θέλω να ξεκαθαρίσω τι γίνεται σε κάθε χώρα. Θα ξεκινήσω από τα του οίκου μου. Με επαγγελματισμό θα εξετάσω τα της χώρας μου. Όπου υπάρχουν παραλήψεις, προβλήματα, θα πρέπει να το παραδεχτούμε. Με την αποδοχή μπορεί να προχωρήσει κανείς. Ιδού λοιπόν κύριε Πρόεδρε. Α, να πω κάτι για το άρθρο 7. Δούλεψα πολύ πάνω σε αυτό το άρθρο όταν ήμουν υπουργό Εξωτερικών. Προέρχεται ουσιαστικά από δική μας πρωτοβουλία. Περιστράφει γύρω από την υπόθεση Χάιντερ στην Αυστρία. Και έτσι άρθηκε η τελευταία επιφύλαξη με την τροποποίηση του άρθρου 7 Ποιο είναι το πρόβλημα τα άρθρο 7. Δεν είναι εύκολο να πετύχει κανείς ειδική πλειοψηφία για να το εφαρμόσει το άρθρο 7. Τούτων λεχθέντων υπάρχει. Είναι ένα μέσο, ένα εργαλείο. Δεν θεωρώ ότι είναι πυρηνική βόμβα. Θεωρώ ότι είναι ένα εργαλείο ως εθεσπίστη και ήταν στόχος, ως εθεσπίστη μέσω της συνθήκης υποχρεώνει διάλογο με την συγκεκριμένη χώρα αυτό το άθρο. Μπορούμε να κάνουμε σύγκριση και με το κοτονού άρθρο 96 και 8 του Κοτονού. Όταν υπάρχει σύγκρουση, πρόβλημα μια χώρα, αυτομάτως ε, υπάρχει υποχρέωση διαλόγου μεταξύ εταίρων. Μοιάζει αυτή η περίπτωση. Το άρθρο 7 δεν είναι ε, μάταιο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί αν υπάρξει πολιτική βούληση. Αυτά. Κατά λοιπά, προφανώς, θα ακούσω προσεκτικά τους συναδέλφους, τις ομάδες και θα προσπαθήσω συνεκτικά να συμπεριλάβω στο κείμενο που θα μεταλλάσσετε τις ιδέες. Θέλουμε να προστατεύσουμε τις αξίες μας, να τις παγιώσουμε και να τις επικαιροποιήσουμε. Ευχαριστώ κύριε Μισελ. Λοιπόν, η τελευταία αυτή παρέμβαση να ανακοινώσω την παρουσίαση σε δύο εκθέσεις που θα γίνει στις 30 Σεπτεμβρίου. 30 Σεπτεμβρίου. Ευχαριστούμε τους συμμετέχοντες στη συζήτηση. Ευχαριστούμε και τον κύριο Μόρτεν Ζέρομ, τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Κύριε Μόρτεν Ζέρομ. Και στις 12 ανακοινώθηκε ότι θα διεξαχθεί κοινή συνεδρίαση Λίβε Γιούρι Αύκο διότι θα ασχοληθούμε με το πρόγραμμα της Στοκχόλμης, είναι μια κοινή έκθεση που συντάσαμε οι συνεισηγητέ, ο υποφαινόμενο εκ μέρου τη Λίμπε, ο κ. Κάρλο Καζίνη εκ μέρου τη ΑΦΚΟ και ο Λουίτζι Μπερλιγκουέρ εκ μέρου τη Γιούρι. στι 12 θα διεξαχθεί η συνεδρίαση. Πρέπει μέχρι τότε να υποδεχθούμε και άλλα μέλη που θα έρθουν, να το έχουμε υπόψη μας, για να εξετάσουμε το σημείο 18 και το 19 κοινή συζήτηση που αφορά τη συμφωνία με την Αρμενία, διευκόλυ... απλούστευση έκδοση θεωρήσεων και επανεισδοχή ατόμων που διαμένουν χωρίς άδεια και είναι σχετικά τα δύο αυτά θέματα. Έχουμε τον ίδιο συγκητή, ήτη, την κυρία Έντιτ Μπάουερ. Της δίνουμε το λόγο λοιπόν και για τα δύο ζητήματα να σας υπενθυμίσω ότι δεν είναι η πρώτη φορά που συζητούμε τα ζητήματα αυτά. Θα καθορίσουν προθεσμία για τροπολογίες αφού ακούσουμε την εισηγήτρια και τους κοιόδης εισηγητές και πρώτα το λόγο τον έχει η εισηγήτρια κυρία Μπάουερ. Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι σύντομη μια και δεν έχουμε πολύ χρόνο. η ανατολική γειτονία έχει ένα νέο μέσο για να ασκεί από εδώ και μπρος την πολιτική της. Η διεύρυνση γιατί η εμβάθυνση της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ένταξης είναι ο στόχος τώρα με την Γεωργία, την Μολδαβία, το Αζερβαϊτζάν, την Αρμενία. Πιστεύω πως έτσι θα συσφίξουμε περισσότερο τις ε, σχέσεις μας και θα γνωρίσουμε ένα τον άλλον καλύτερα. Το Σεπτέμβριο του 2012 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άρχισε τις διαπραγματεύσεις για την συμφωνία αυτή και στις 17 Σεπτεμβρίου υπογράφηκε η συμφωνία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όμως πρέπει να εγκρίνει την συμφωνία. Ήδη εννέα χώρες, δέκα μάλιστα, έχει, έχουν συμφωνήσει για χαλάρωση των κανόνων ε, για έκδοση θεώρησης ε, για τις χώρες του Καυκάσου, της Αιγεωργίας ε, συμπεριλαμβανομένης και με το Αζερβαϊτζάν οι διαπραγματεύσεις προχωράνε. Τώρα τι γίνεται με το Αζερβαϊτζάν. οι διαπραγματεύσεις εξελίσσονται θετικά. Υπήρξε ένα πρόβλημα με το Αζερβαϊτζάν. Υπήρχε λοιπόν ένα πρόβλημα με το σύμφωνο έκδοσης. Τα προβλήματα όμως αυτά παραμερίστηκαν. Γι' αυτό λοιπόν και θεωρούμε πως είναι πολύ σημαντικό ήδη στη συνοπτική αιτιολόγηση να αναφέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να επιταχύνει την διαδικασία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Ίσως κάτι τελευταίο, κάτι το οποίο απασχολεί την Ευρωπαϊκή Εξωτερικών Υποθέσεων, να πω ότι στηρίζουμε το έργο της και να... Να σας πω ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε πλέον το κείμενο, διότι η αλλαγές που θα προταθούν πρέπει να είναι μόνο για το έγγραφο που έχουμε εμείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ας ακούσουμε τώρα και τους κύριους ηγητές. Κυρία Κιγιώμη. Ναι, εν συντομία. Καταρχήν λυπάμαι που οι σκιώδεις δεν συναντήθηκαν να συζητήσουν το θέμα αυτό, αναγνωρίζοντας βέβαια ότι το θέμα δεν είναι ε, και μείζον. Έτσι κι αλλιώς ε, έχουμε και περιορισμένο περιθώριο ε, ε, παρέμβαση σε μια και το 2013 υπογράφηκαν οι συμφωνίες και για την απελευθέρωση της, ε, των θεωρήσεων και για την επανεισδοχή. Πρόσφατα ξεκίνησε η στοχευμένη πρωτοβουλία για την Αρμενία που έχει ως στόχο την ενίσχυση των, της ικανότητας των αρμενικών αρχών να χειριστούν την ε, μετανάστευση. Είναι καλό λοιπόν να περιγράψουμε το σύνολο του πλαισίου μέσα στο οποίο κινούμαστε. Θα πρέπει να υποστηρίξουμε λοιπόν την απελευθέρωση την, της έκδοσης θεωρήσεων με χώρα όπως η Αρμενία που έχουν ιστορικούς δεσμούς μαζί μας. Ε, δεν συμφωνώ πλήρως με την εισηγήτρια για τα όσα λέει ότι θα πρέπει να ε, κάνουμε προσπάθειες να υπογράψουμε παρόμοιες συμφωνίες με το Αζερβαϊτζάν. Θα είμαστε, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί γιατί υπάρχουν διαφορές προβληματική είναι τελείως διαφορετική, ιδιαίτερα σε θέματα μετανάστευση. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη Συμφωνία πανεισδοχή. Μεταξύ των προτεραιοτήτων της ομάδας μας είναι τα κράτη-μέλη να εγγυώνται στους υπηκούς τρίτων χωρών που βρίσκονται στην επικράτειά τους τη δυνατότητα να ζητήσουν ε, διεθνή προστασία αν το επιθυμούν και υπό την ε, αίρεση της αρχής της ε, μη επαναπρόθεσης. Τέλος, να υποφελθώ τι ευκαιρία αυτή προκειμένου να ε, ρωτήσω την Κομισιόν τι γίνονται με τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει κατά την υπογραφή της συμφωνίας επανεισδοχής του Πακιστάν πριν από, με το Πακιστάν πριν από τρία χρόνια, το 2010, το Σεπτέμβριο 2010. Είχε δεσμευθεί ε, να υποβάλει εκθέσεις στο κοινοβούλιο σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της, των συμφωνιών επανεισδοχής. Τι γίνονται με αυτές τις δεσμεύσει. Η κυρία Στανόκα. Όχι, ο κύριος Σίλτσεφ θα λάβει πρώτο το λόγο. Τον... Έχετε ζητήσει το λόγο, σωστά. Ωραία, κυρία Στάνοκα, πρώτα και μετά κύριο Σίλτσεφ. Συγχαίρω την κυρία Μπάουερ για τη δουλειά που έκανα, για την προετοιμασία της έκθεσης, σαν ομάδα των Πρασίνων. Ξέρετε ποια είναι η θέση μας. Έχουμε επιφυλάξεις όσον αφορά τις συμφωνίες επανεισδοχής, συγκεκριμένα με χώρες όπου υπάρχουν περιφέρειες με αβεβαιότητα στον αφορά το καθεστώς που τις διέπει Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν κάποιες διαδικασίες επανεισδοχής με τέτοιες χώρες και είχαμε αντιρρήσεις. Και στην περίπτωση άλλων χωρών της περιοχής του Καυκάσου και σε άλλα μέρη του κόσμου. Έτσι και εδώ έχουμε επιφύλαξη. Όσον αφορά τη διευκόλυνση θεωρήσεων, πάντα είμαστε υπέρ Είμαστε υπέρ ελεύθερης διακίνησης των ανθρώπων και υποστηρίζουμε αυτή την ιδέα. Όμως, λαμβάνοντας υπόψη την πολύ ευαίσθητη κατάσταση όσον αφορά παρόμοιες συμφωνίες που εξετάζονται με το Αζερμπαϊτζάν θέλουμε να υποστηρίξουμε τη διευκόλυνση θεωρήσεων και τη σχετική συμφωνία ως έχει με την Αρμενία αλλά να βάλουμε μία φράση, να προσθέσουμε. Να λέμε ότι αυτή η συμφωνία τίθεται σε ισχύ παράλληλα με παρόμοια συμφωνία με το Αζερμπαϊτζάν. Αυτό μπορούμε να το υποβάλουμε, να υποβάλουμε μια τέτοια τροπολογία, μια τέτοια πρόταση να προσθεθεί. Αυτό θα κάνουμε και έτσι προτείνουμε να λυθεί το πολύ ευαίσθητο πρόβλημα, να υπάρχουν καλές σχέσεις δηλαδή με όλου τους γειτονές μας της ανατολική Ευρώπης. Και πρέπει να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση στις εργασίες μας. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Ήλτσεφ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εκ μέρους της Άλτε θέλω να εκφράσω υποστήριξη για τα δύο αυτά ζητήματα. Εκτιμώ το έργο της εισηγήτριας της κυρίας Μπάουερ. Με ακρίβεια κινήθηκε και εγκαίρος. Η υπογραφή αυτών των συμφωνιών για την επανεισδοχή και για τη διευκόλυνση των θεωρήσεων είναι κάτι που δημιουργεί πιθανότητες για περαιτέρω και συνθήκες για περαιτέρω μεταρρυθμίσεις. Και η Αρμενία Αξίζει με τέτοια χειρονομία πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διότι η Αρμενία έκανε πολλές μεταρρυθμίσεις ε, πρόσφατα και εφάρμοσε κάποιες βασικές νομοθεσίες για να αποκριθεί στις προσδοκίες ευρωπαϊκές με επάρκεια. Επιτυχώ εφάρμοσε μεταρρυθμίσεις, χωρί δισταγμό μπορούμε να υποστηρίξουμε τι δύο εκθέσει και θα πρέπει να ολοκληρωθούν αυτέ οι δύο συμφωνίε. Θυμάμαι αυτά που είπε επίτροπο, η Επίτροπο κυρία Μάλστρομ είπε ότι αυτές οι δύο συμφωνίες είναι απτά αποτελέσματα της ανατολικής γειτονικής σχέσεως και θα προωθήσουν τη διάδραση μεταξύ πολιτών Ευρωπαϊκής Ενώσεως και Αρμενίας και θα ενισχυθεί η συνεργασία μας στην καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης. Και μπορώ να προσθέσω ότι αυτό το γεγονός θα ενθαρρύνει επίσης και τους γείτονες της Αρμενίας, συμπεριλαμβανομένου του Αζερβαϊτζάν, να προχωρήσουν πέρα της συνήθους ερμηνείας που ισχύει σε αυτές τις περιπτώσεις Δηλαδή, ελπίζουμε ότι το γειτονικό Αζερμπαϊτζάν θα προωθήσει κάποιες διαδικασίες, ούτως ώστε τέτοια ανάλογη εξέλιξη να αναμένεται που θα τη και στις προσδοκίες του Αζερμπαϊτζάν. Μπορούμε επίσης να πούμε ότι η, Γεωργία, ή μάλλον η Αρμενία προστίθεται σε μια μεγάλη ομάδα χωρών που απολαμβάνουν τα ωφέλη αυτών των καθεστώτων. Χώρες όπως η Μόδοβα, το Μαυροβούνιο, η Ρωσία, η Σερβία, η Ουκρανία και η Γεωργία. Ας πούμε ότι αυτές οι πολιτικές είναι μια λογική ε, προσπάθεια εξορρόπησης ανάγκης εσωτερικής, για εσωτερική ασφάλεια και εξωτερική σταθεροποίηση στη γειτονιά της Ευρώπης. Άρα αυτό σημαίνει ότι κινούμαστε προς σωστή κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Εκτός μικροφώνου ο Πρόεδρος. Μάλλον ρωτάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Συμβούλιο ε, επιθυμούν να σχολιάσουν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ορίστε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, εντάχει, σε ό,τι αφορά τη συμφωνία πανεσδοχής με την Αρμενία ιδιαίτερα, αποτελεί τμήμα ενό πακέτου που συνάπτουμε με την Αρμενία στο πλαίσιο της ανατολικής εταιρικής σχέσης όπως είπε ο εισηγητής. Κινητικότητα σε ένα ασφαλές περιβάλλον σημαίνει ότι η Συμφωνία Απελευθέρωσης Θεωρήσεων ε, ακολουθείται, συνοδεύεται από μια ε, συμφωνία διότι η αυξημένη κινητικότητα οδηγεί σε αυξημένους κινδύνους ε, μετανάστευσης. Τώρα, μια-δυο παρατηρήσεις σχετικά με το θέμα της μεταχείρισης ε, των ετούντων άσυλο ή ετούντων διεθνούς προστασίας στο πλαίσιο της Συμφωνίας Επανεισδοχής. Η ετουντων διεθνης προστασιας στο Επανεισδοχής ε, υφίσταται ε, με την επιφύλαξη της συνθήκης για την μεταχείριση των ετούντων άσυλο. Παίρνουμε πάρα πολύ στα σοβαρά τις υποχρεώσεις μας. Το 2011 η Κομισιόν υπέβαλε μια ανακοίνωση που περιελάμβανε ένα αριθμό συστάσεων για την ενίσχυση της προστασίας των θεμελιών δικαιωμάτων στο πλαίσιο των συμφωνίων επανειστοχής, αυτές οι συστάσεις οδήγησαν σε νέες διατάξεις, οι οποίες βλέπετε για πρώτη φορά σε αυτή την συμφωνία επανειστοχής με την Αρμενία, ιδιαίτερα σε ένα νέο άρθρο 2, το οποίο προστίθεται και εξασφαλίζει το σεβασμό των θεμελιών δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επανειστοχής, καθώς επίσης και το σεβασμό των ατόμων τα οποία επιστρέφονται μέσω μιας τέτοιας συμφωνίας επανεισδοχής. Επίσης, ε, δίδεται προτεραιότητα στην εκούσια επιστροφή. Ε, θα δείτε και μια άλλη ε, καινοτομία. Προστίθεται μια ρήτρα αναστολής που προβλέπει πως αν υφίστανται μακρόχρονα και τακτικά προβλήματα ε, ε, ε, παραβίαση θεμελιών δικαιωμάτων, τότε υπάρχει δυνατότητα αναστολή. Για την Αρμενία δεν βλέπουμε τέτοιο θέμα. Είναι συμβαλόμενο μέρο σε πολλέ διεθνεί συμφωνίε και στην Συμφωνία Επανεισδοχή στην οποία αναφέρατε. Ευχαριστώ. Άλλα σχόλια. Ο πλευρά Προεδρία, όχι. Επιστρέφουμε στην συγκίτρια την κυρία Μπάουερ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για όλα τα σχόλια. Θα έχουμε χρόνο να συναντηθούμε πρώτα με τους κοιόδες ηγητές, να τα συζητήσουμε πρωτού οδηγηθούμε στο τελικό έγγραφο. Ξέρετε όλοι ότι όταν έρχονται στο Κοινοβούλιο διαφορετικές προτάσεις, πολλές φορές έχουμε δυσκολίες και καθυστερήσεις. Στην περίπτωση του Αζερμπαϊτζάν η καθυστέρηση οφειλόταν στο ότι το Αζερμπαϊτζάν δεν έδειξε πολιτική θέληση ως προς την συμφωνία για τις θεωρήσεις. Δεν έχει αλλάξει αυτή η κατάσταση μέχρι τώρα. Επίσης, είχαμε πάρα πολλές αιτήσει για άσυλο από άτομα από το Αζερβαϊτζάν και αυτή η κατάσταση άλλαξε. Γι' αυτό πιστεύω πως έχει έρθει η ώρα να ασχοληθούμε σοβαρά με το θέμα αυτό που συνδέεται και με τη συμφωνία με την Αρμενία. Όπως είπαν και ορισμένοι συνάδελφοι, ο κύριος Σίλτσεφ για παράδειγμα, δεν υπάρχει λόγος να μην δώσουμε τη συγκατάθεσή μας για να τέθει σε ισχύ η συμφωνία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Μπάουερ. Αυτά προς το παρόν. Να σας ανακοινώσω μόνο ότι η προθεσμία για τροπολογίες είναι η 15η Ιουλίου. Σας υπενθυμίζω ότι σε περίπτωση διεθνούς συμφωνίας θα γίνονται δεκτές μόνο τροπολογίες επί της διαδικασίας, έτσι ώστε η ψηφοφορία να διεξαχθεί στην συνεδρίαση μας στις 16 και 17 Σεπτεμβρίου. Σας ευχαριστώ όλους. Και τώρα θα έχουμε χρόνο να προετοιμαστούμε για την κοινή συνεδρίαση με τις Επιτροπές Συνταγματικών Υποθέσεων και Νομικών Υποθέσεων για να συζητήσουμε το πρόγραμμα της Στοκχόλμης. Πέντε λεπτά διάλειμμα και μετά αρχίζουμε. Ευχαριστώ.